Morning, dear, dear colleagues. I would like... Καλημέρα. Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Πριν καλωσορίσουμε τον Μάριο Σεντένο, τον πρόεδρο του Eurogroup, να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα έγγραφα της συνεδρίασης. Ε, θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχετε τα συνήθεια έγγραφα μπροστά σας. Αυτό κατόπιν του email της 6ης Δεκεμβρίου που τροποποίησε την σχετική πολιτική για να συνεισφέρουμε στην μείωση των εκπομπών οπότε ο κανόνας είναι ότι μόνο οι βουλευτές που έχουν ζητήσει τα έγγραφα έχουν όπως βλέπω κάποιους μπροστά μου να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσετε ε, να ζητήσετε ή να ζητήσετε να μην λαμβάνετε τα έγγραφα οπότε μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την γραμματεία Σύνοψη των αποφάσεων των συντονιστών στις 23 Ιανουαρίου έχουμε ορισμό, απλοποίηση κάποιων κανόνων στο σύστημα το φορολογικό σοσιαλδημοκράτες, διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ ΓΚΟΕ, τροποποιημένη πρόταση για έναν κανονισμό για την ενισχυμένη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ πάει στο ECR, κοινό σύστημα ΦΠΑ σε σχέση με κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές πάει στο Προεδρείο, ύψος ΦΠΑ σοσιαλδημοκράτες, κοινό σύστημα ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις ΕΛΚ, προληπτική εποπτεία επενδυτικών εταιριών ΕΛΚ, προληπτικές απαιτήσει επενδυτικών εταιριών ΕΛΚ, προπολογισμό 2019, όλα τα τμήματα πάει στο Προεδρείο Brexit. Οι συντονιστές συζήτησαν και συμφώνησαν τις περαιτέρω πτυχές της μεθόδου εργασίας. Αντιπροσωπεία στην Γαλλία 12 έως 14 Φεβρουαρίου 2018. και ήταν πολύ επιτυχημένη η αποστολή. Δημόσιες ακροάσεις αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά με κάποιους προσκεκλημένους. Μετά έχουμε τους μελλοντικού διορισμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμφωνήσαμε με τα βήματα που πρέπει να γίνουν και θα τα συζητήσουμε Δευτέρα και Τρίτη. Μετά οικονομική διακυβέρνηση. Αποφασίσαμε τις ημερομηνίες για την αποστολή στην Αθήνα και το τι θα κάνουμε για την εποπτεία μετά το πρόγραμμα, για τις χώρες που είναι σε πρόγραμμα για τις μελλοντικέ συναντήσεις ε, της ομάδας εργασίας ε, για την ε, δημοσιονομική βοήθεια, για τους διορισμούς στην ΕΖΑΚ, για το ελεγκτικό συνέδριο, τις ειδικέ εκθέσεις και για ζητήματα που θα συζητηθούν όπως παραδείγματος χάρη το σχέδιο Γιούνκερ αν έχει προσελκύσει επιπρόσθετες επενδύσεις, αξιολόγηση των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων, εξέταση των πράξεων κάτω εξουσιοδότηση, ενημέρωση μαζί με τον πρόεδρο του, την πρόεδρο του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας. Αυτά σας ευχαριστώ. Έχουμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 11 η Ιανουαρίου και την ημερήσια διάταξη και τέλος καλωσορίζω τον πρόεδρο του Eurogroup τον Μάριο Σεντένο για τον τακτικό οικονομικό διάλογο που έχουμε θεωρώ ότι έχουμε εδώ πέρα ένα θετικό μήνυμα το ότι εμφανιστήκατε χτες στην διακοινοβουλευτική διάσκεψη με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και σήμερα είστε εδώ στην Επιτροπή μας για την πρώτο οικονομικό σας διάλογο με βάση τον κανονισμό 1466 του 97 οπότε ορίζουμε την ευκαιρία να ξεκινήσει ένας ε, τακτικός διάλογος μαζί σας και αναμένουμε μια ενισχυμένη συνεργασία και διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Eurogroup λαμβάνοντας ιδιαίτερος υπόψη την φάση την οποία περνάμε είπαμε ότι έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για να ληφθούν κάποια αποφασιστικά βήματα για να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική μας Ένωση η Επιτροπή μας επίσης ε, θα ήθελε να μας πείτε κάποια πράγματα για τα αποτελέσματα του Eurogroup της Δευτέρας, ειδικά για την Ελλάδα και για το τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας ε, και ξέρω πως υπήρχε και μια έντονη συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση. Πολλά πράγματα λοιπόν να συζητήσουμε. Λοιπόν, Μάριο, έχετε τον λόγο. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Είναι μεγάλη μου ικανοποίηση να βρίσκομαι εδώ στην ε, Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πρώτο οικονομικό διάλογο και θεωρώ ότι ο ρόλος μου για η δημοκρατική λογοδοσία είναι πάρα πολύ σοβαρό και οπότε και εγώ θα έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ για να συζητούμε τι οικονομικέ εξελίξει. Και θα αρχίσουμε δυο λόγια όσον αφορά την οικονομική συγκυρία και στη συνέχεια να δούμε ποιο είναι το, το οποίο που αφορά το έργο μα, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα των εθνικών πολιτικών, επίση να δούμε τι γίνεται με την ε, Οικονομική Νομισματική Ένωση και θα ολοκληρώσουμε κάποια ενημέρωση όσον αφορά το πρόγραμμα προσαρμογής της ε, Ελλάδος. Τώρα όσον αφορά την οικονομική συγκυρία βλέπουμε τώρα την ρόδινη πλευρά του οικονομικού κύκλου και αυτό δεν ε, συμβαίνει τυχαία. Αυτό ε, είναι συνέχεια σκληρής δουλειάς και η οικονομία μας βλέπουμε ότι έχει γίνει πρωτοπόρα στην ε, παγκόσμια οικονομία και μπορούμε να θυμούμε ότι έχουν περάσει 19 επιτυχή τρίμηνα όσον αφορά κάποια ευρεία βάσεις ε, αυξανόμενη ανάπτυξη και αύξηση του ΑΕΠ. Και όλα αυτά λόγω των μεταρρυθμίσεων που κάναμε και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αντίδραση προς την κρίση ίσως ήταν βραδία Όντω ισχύει αυτό, ιδίω όσον αφορά την απασχόληση αλλά και τι επενδύσει. Όμω, σιγά σιγά μπορέσαμε τι ανισορροπίε να τι ε, διορθώσουμε και μπορέσαμε να συγκροτήσουμε την αρχιτεκτονική του ευρώ. Και τα προγνωστικά λένε ότι πρόκειται τις επόμενες χρονιέ να χυστεί ο θετικός ρυθμό ανάπτυξη και αυτό ε, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να υποχωρούν οι ανισορροπίες. Έχουμε επομένως θετικές ροές στην οικονομία μας που είναι το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων και επίσης συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις ακόμα και τώρα. Και επομένω γι' αυτό έχουμε θετικού ρυθμού όσον αφορά την απασχόληση, επίση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και επίση ε, η εξωτερική μα οικονομική πολιτική είναι υγιή. Οπότε τώρα προσπαθούμε να έχουμε μια τέτοια βιώσιμη ανάπτυξη και θεωρούμε ότι ε, ό,τι μας κλωδόδησε η κρίση πρόκειται να αρθεί μέσω αυτής της ε, θετικής οικονομικής τάσης. Θα πρέπει επίσης τα fundamentals να τα βελτιώσουμε ακόμη και να προχωρήσουμε σε περισσότερη ανάπτυξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός δηλαδή ο ενάρετος κύκλος να συνεχιστεί. Οπότε τώρα ερχόμαστε στο ζήτημα του πώληση μίξ που το οποίο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο τόσο ώστε η ευρωζώνη και οι οικονομίες της να είναι διορθωτικά πιο δυνατέ, θα πρέπει να έχουμε ισόρροπη ανάπτυξη και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται ε, να υπάρχουν κάποιες προσεκτικά σχεδιασμένες εθνικές πολιτικές με τους εξής στόχους να δούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται ούτως ώστε να απορροφήσουμε τις ε, διαταραχές από ό,τι προηγήθηκε και τώρα επομένως θα, πρέπει να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε με δημοσιονομικά μέτρα να ξεπεράσουμε τις ε, Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να συνεχίσει να εφαρμόζει τους σχετικούς ε, κανόνες με λογική. Επομένω χρειάζονται κάποιες δημοσιονομικές πολιτικές ε, στεγανές, αλλά δεν αρκούν αυτές για να πετύχει το οικονομικό μοντέλο. Θα πρέπει να μπορέσουμε επίσης να συνεχιστεί αυτή η αναπτυξιακή τάση, ακόμα και σε χειρότερη συγκυρία. Χρειάζεται κάποια ε, αντοχή για όλες τις χώρες, γιατί πολλές φορές ε, χρειάζεται πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, και να στο πιο από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Επομένω, θα συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στην ανταγωνιστικότητα, ούτε ώστε να έχουμε υψηλής ποιότητας επενδύσεις και να αποτελέσουν αυτό, αυτές τις προτεραιότητές μας. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρωζώνη τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά πολλά χρόνια τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ιδίω κατά την κρίση και αμέσως μετά. Οπότε χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες με δεδομένη με δεδομένο το, το περιβάλλον σχετικά με τα επιτόκια. Οπότε θα πρέπει η οικονομία να έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί στις ε, προκλήσεις της ε, παγκοσμιοποίησης. Οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε περιβάλλον τόσο ώστε να μπορούν να, να καινοτομήσουν και να επενδύσουν οι επιχειρήσεις μας. Επίσης θα πρέπει η απασχόληση να είναι πιο ελκυστική και θα πρέπει επίσης να αποδίδει πλάς παραγωγικότητα. Επίσης είναι και το θέμα κάποιες δίκαιες φορολογίας, παιδείας και κατάρτισης επαγγελματικής. Δηλαδή τέτοια πρόοδο θέλουμε ώστε να μην αφήνει κανένα να παίξουν έναν οικονομικό μοντέλο που να ωφελεί όλες τις χώρες. Οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας που ακόμα τις έχουμε στη μεγάλη μας ενιαία αγορά. Το δε Eurogroup κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συνεχίσει να ε, παίζει ε, έναν ρόλο καταλήτη θετικό για όλα αυτά και κυρίω από τότε που η... Ε, είναι δεδομένο ότι είναι αλληλένδετες οι οικονομίες. Οπότε χρειάζονται κάποιες πρωτοβουλίες και απλώς δημοσιονομικής ε, οπότε θα πρέπει αυτές μας οι πολιτικές να έχουν επιπτώσεις και ε, διασυνοριακά. Όλα αυτά πολύ καλά στο χαρτί, αλλά για να αποδώσουν θα πρέπει να διαχειριστούμε τις προσδοκίες μας και θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι στη δημόρφωση πολιτική να ακολουθούν. Γι' αυτό πάντοτε σαν βούληση δεν υπάρχει στην πολιτική ζήμωση. Ξέρουμε από την πείρα μας ότι κάποιες πολιτικές ε, θα φέρουν την ανάπτυξη που θέλουμε. Για να δούμε τώρα και να στραφούμε στο πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε την ε, Νομισματική Ένωση και είναι ευθύνη μας Παρασκευή για το μέλλον αλλά είναι συλλογική αυτή η ευθύνη όσον αφορά την Ένωση. Θα πρέπει μενος η Νομισματική Ένωση να αποκτήσει βάθος. Και χθε είπα τις απόψεις μου σε εκείνη τη διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό εξάμεινο στα πλαίσια της κοινοβουλευτική ε, ομάδας και είπαμε ότι θα πρέπει να δουλέψει σκληρά η Οικονομικών και τον Ιούνιο η Ελληνική Κανονική Κυβέρνηση να λάβουν τι ανάλογε αποφάσει, να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και την ε, περαιτέρω ολοκλήρωση του ESM. Και αν θέλουμε όλα αυτά να αποδώσουν, θα πρέπει να εστιαστούμε στα θέματα ουσία. Ο χάρτη προς το 2016 είναι η βάση μας, γιατί δεν αρχίζουμε από το 0. Τον ε, Ιούνιο χρειάζεται να έχουμε κάποιους σαφείς, ξεκάθαρους στόχους και δεν τελειώνει το θέμα εδώ. Είναι ε, η αρχή μιας νέας φάσης ε, υλοποίησης και θα πρέπει να διευνήσουμε και άλλες λύσεις κοινή, κοινή δημοσιονομική δυνατότητα, κοινού κανόνε. Γιατί δεν μπορούμε βέβαια να προδικάσουμε το που θα καταλήξουν οι Υπουργοί Οικονομικών ή οι αρχηγοί κρατών στι ε, συναντήσει κορυφή του. Αλλά θεωρούμε ότι θα καταλήξουν σε κάποιε αποφάσει μεστέ νοήματο και φυσικά υπάρχει η πολιτική βούληση. Μπορούμε έτσι να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αποφασει που παρουσιάζεται και ήδη ε, έχουμε κοινέ απόψει οι οποίες μπορεί να είναι αφετηρία. Και όλα αυτά θα έχουν σκοπό το ότι θα πρέπει η Ευρωζώνη να αποκτήσει περισσότερη ανθεκτικότητα και έτσι θα εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα αναλυφθούν οι ίδιοι κίνδυνοι όπως και στο παρελθόν ο τότε που το ευρώ δεν ήταν έτοιμο να αντισταθεί στην ε, κρίση. Εάν ισχυροποιήσουμε το ευρώ ε, έτσι ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο δώρο στους πολίτες μας και θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εμπιστοσύνη και όπως ανέφερα χθε στο κοινοβούλιο εδώ δεν είναι αυτός σκοπός το ευρώ είναι μέσο προς επίτευξη των σκόπων μας Τώρα για την Ελλάδα. Από την αρχή τη δεκαετία είχαμε αυτά τα προβλήματα μικρή προσαρμογή στην Ελλάδα και αυτό ήταν πάγιο θέμα ζήτηση στο Eurogroup και όσον αφορά επίση τι συναντήσεις, τους οικονομικούς διαλόγους με τους προκατόχου μου και ήταν δύσκολη αυτή η διαδρομή και φυσικά κυρίω δύσκολη για τους ε, Έλληνε πολίτε. Ε, αυτοί θα έπρεπε να περάσουν τα πιο δύσκολα. Πάντως ε, τώρα τα μαντάτα είναι ενθαρρυντικά και με τα στοιχεία που έχουμε αυτό προκύπτει ότι η, ευρωπαϊκή, η ελληνική οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη πέρσι και υπάρχει τώρα πρόσβαση στις αγορές το περιβάλλον δείχνει θετικό και τον Ιανουάριο το Eurogroup κατέληξε σε κάποια πολιτική συμφωνία όσον αφορά την τρίτη αξιολόγηση. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά και οι ελληνικές αρχές τώρα ουσιαστικά ε, εφαρμόζουν ό,τι εκκρεμούσε. Επομένως φαίνεται θετική η ατμόσφαιρα. Και άπαξ και ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, ο ΕΣΥΜ μπορεί να προβεί σε άλλη μια εκταμείευση και ε, ούτως ώστε να υπάρξει ε, αυτού του είδους ε, η χρηματοοικονομική ροή που χρειάζεται η Ελλάδα. Οπότε και θα μπορεί να βγει από το πρόγραμμα του ESM η Ελλάδα όπως προβλέπεται να γίνει τον Αύγουστο φέτος, τους αμέσως επόμενους μήνες. Το Eurogroup πρόκειται να εξετάσει το πώς θα επιστρέψει η Ελλάδα σε κάποιο βιώσιμη πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές και χρειάζεται βέβαια τεχνική εργασία και κάποια μέτρα σε σχέση με το χρέος ομόφωνα τον Ιούνιο από αυτού συνεφώνησε το Eurogroup και θα ληφθεί αυτή η απόφαση περί το τέλος του προγράμματος μόλις υπάρχει μια ενημέρωση πλήρης <clears throat> και όταν έχουν γίνει σχετικές αναλύσεις. Τώρα όσον αφορά το μέλλον θα πρέπει όλα αυτά να τα εστερνιστεί κανείς για να πετύχουν και ξέρω προσωπική εμπειρία ως Υπουργός Οικονομικών της χώρας μου. Χρειάζεται να υπάρχει τέτοιου είδους ενστερνισμός των ε, αποφάσεων της στρατηγικής ώστε τα καλά αποτελέσματα και επιδόσεις να μην πάνε χαμένα. Η Ελλάδα θεωρούμε ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα σοβαρά, ετοιμάζει η κυβέρνηση αυτή τη μακρόπνη στρατηγική την οποία θα παρουσιάσει στο Eurogroup και αυτή η στρατηγική ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντική ούτως ώστε να σχηματιστεί, να διαμορφωθεί το πλαίσιο για τη συνέχεια και επομένως έτσι να είναι ισότιμη η χώρα με τους Ευρωπαίους εταίρους της και η κρίση να αποτελέσει ένα ε, θέμα του παρελθόντος. Και εμείς περιμένουμε πώς και πώς αυτό να γίνει πραγματικότητα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο για τα σημαντικά αυτά σχόλια. Πράγματι, εχθές είχαμε μια εξαιρετική ανταλλαγή με τον Υπουργό Οικονομικών. Σημειώσαμε την πρόοδο που έχει γίνει. Είχαμε μια συνολικά θετική αξιολόγηση της ε, δουλειάς που έχει γίνει και από τις δύο πλευρές ε, και από την ελληνική κυβέρνηση και από τα θεσμικά όργανα για τον ESM ε για να αναπτυχθεί μια στρατηγική οικονομικής μέγεθυνσης. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά μπορούν να καταλήξουν σε απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα. Θα πάμε τώρα στον κύκλο παρατηρήσεων και ερωτήσεων. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεντένο, Σας καλωσορίζω και εγώ. Χαίρομαι που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, νομίζω ότι εκπροσωπώ όλη την ομάδα του ΕΛΚ όταν λέω ότι χαιρόμαστε για την συνεργασία μαζί σας. Έχω μια ερώτηση που έχει σχέση με την συνεδρίαση του Eurogroup ε, αυτή την εβδομάδα. Ε, εκεί πέρα είπατε ότι Θέλετε ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ταυτάχρονα αποκλείεται μεταφορές ε, κεφαλαίων σε χώρες ε, με ασθενή τραπεζικά συστήματα και ότι ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν οριακές ε, περιπτώσεις και μάλιστα λέγεται ότι το σύστημα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων όταν έχουν υπάρξει υπερτέρω βήματα στο θέμα μείωση του κινδύνου αλλά βεβαίως ε, όποιος ε, λέει το α φίλοι να πει μετά και το Β. Δεν θα πρέπει λοιπόν να καταλήξετε στο Eurogroup σε συγκεκριμένες προτάσεις για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ενίσχυση της ε, κεφαλαιοποίησης ε, για να υπάρξει μια αξιόπιστη και τονίζω την λέξη αξιόπιστη μείωση του κινδύνου και ακριβώς τώρα που είναι καλή θα έλεγα η οικονομική συγκυρία να πείσετε τους συναδέλφους σας να κάνουν ε, κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Μπάλτς για την πολύ σημαντική αυτή ερώτηση επί πολύ σημαντικού θέματος. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί το θεσμικό τοπίο της Τραπεζικής Ένωσης προς το όφελος όλων των συμμετεχόντων και προκειμένου να είναι έτσι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν εμπιστοσύνη στα βήματα που πρέπει να αναλάβουμε και να αποφευθούν οποιασδήποτε οποιαδήποτε αν θέλετε κίνητρα που δεν συνάδουν προς την, κατεύθυνση αυτήν. Είχαμε λοιπόν συμφωνήσει από το 2016 σε μια υλοποίηση μέτρων μειώσεως του κινδύνου τα οποία συζητώνται εδώ και αρκετό καιρό πλέον και εκτιμώ ότι αυτά θα εγκριθούν στην δέσμη μέτρων μείωσης του κινδύνου που είναι υποσυζήτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός προκειμένου να περιορίσουμε τον κίνδυνο στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εξέλιξη των δικτών που έχουμε μέχρι στιγμής είναι και απόρρια των μέτρων που έχουν ληφθεί ώστε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας και βέβαια ευρεία δέσμη μέτρων έχει ήδη ληφθεί όλες οι οδηγίες CRR, CRD, 4, BRD, η υλοποίηση του ενιαίου μηχανισμού επιτήρησης όλα αυτά και άλλα ενισχύουν την αξιοπιστία του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι αλήθεια ότι κάποιες χώρες, όλες οι χώρες υποφέρουν από την κρίση, αλλά είχαν, κάποιες χώρες είχαν πληγεί ιδιαίτερα. Και κάποιοι εθνικοί τομείς, τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί, αντιμετωπίζουν μια παράδοση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και η μείωση της πίεσης που αναφέρατε είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι αυτό το παρελθόν, αυτή η παράδοση είναι κάτι που θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Και ένας δείκτης τον οποίο ήθελα να αναφερθώ ήταν ακριβώς στο πλαίσιο του μηχανισμού επιτήρησης για όλες τις τράπεζες όλες οι τράπεζες που επιτηρούνται έχουν ξεπεράσει τα περιθώρια βαθμολόγησης, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που τους είχαν τοποθετηθεί, επίδοσης. Αυτό είναι η βασική μου δουλειά ως πρόεδρος του Eurogroup, δηλαδή παρατηρούμε την εξέλιξη αυτή. Είχαμε το 25% της μείωσης το 2017 και μισός ποσοστιαίος βαθμός ε, ήδη στους πρώτους βαθμούς του 2018. Επομένως δηλαδή η τάση είναι πράγματι ουσιαστική, δεν είναι αμεληταία. Τώρα, ο κύριος Περέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Θεντένο να τον καλωσορίσω θερμά από πλευράς ε, της ομάδας S&D και να εκφράσω και μια ικανοποίηση ως Πορτογάλος και ως Ευρωπαίος. Ως Πορτογάλος πολίτης διότι έως και πρόσφατα συζητούνται κυρώσεις κατά της χώρας μου. Η εκλογή σας ε, στη θέση του Προέδρου είναι ένα, μια απόρρεια, ένα δείγμα της σοβαρή δουλειά που είχατε κάνει και ω Υπουργό Οικονομίας. Αλλά και ως Ευρωπαίος εκφράζω την ικανοποίησή μου, διότι η εκλογή σας είναι ένα σημάδι ελπίδας για το μέλλον του ευρώ και της ευρωομάδας. Και βεβαίως πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία των ε, μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης εγώ έχω παρακολουθήσει την διαδικασία των συζητήσεών σας, της εκλογής σας. Ο στόχος της ολοκλήρωσης λοιπόν της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι ουσιοδέστατος, αλλά και η προαγωγή της σύγκλησης. Και η ικανοποίηση, εν πάση περιπτώσει, των προσδιοκίων των πολιτών. Επομένως, αυτός ο στόχος της σύγκλησης, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πόσο σημαντικός είναι. Και επίσης ήθελα να καταλάβω κατά πόσον αυτή η φιλοδοξία της σύγκλησης είναι συμβατή με το μινιμαλιστικό πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί που περιορίζεται στην Τραπεζική Ένωση που δεν έχει ικανότητες να αναλάβει τα δημοσιονομικά του άχθη και με μια εξέλιξη πρόοδο του μηχανισμού σταθερότητας προς ένα νομισματικό ταμείο το οποίο, του οποίου θα έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα ενίσχυση της σταθερότητας στην πραγματικότητα. Και επομένω, με την έννοια αυτή πώς θα υλοποιήσουμε τη φιλοδοξία αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Περέιρα και θα απαντήσω στα πορτογαλικά ε, στην ερώτησή σας. Σας ε, επιβεβαιώνω λοιπόν ότι πράγματι έχουμε πολύ σημαντική φιλοδοξία εκφράσει και έχουμε μία μοναδική ευκαιρία στρατηγική όχι μόνο λόγω του χρονικού σημείου του πολιτικού κύκλου Υπάρχει μια έντονη φιλοδοξία λοιπόν που εκφράζεται και που τροφοδοτείται αν θέλετε και ενισχύεται από αυτόν τον πολιτικό κύκλο στον οποίο αναφέρομαι και τη συγκεκριμένη βεβαίως ε, χρονική στιγμή οικονομικός μιλώντας που ζούμε. Επιθυμούμε όμως και εξακολουθούμε να έχουμε την φιλοδοξία να ενισχύσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Νομίζω ότι έχουμε θετικούς δείκτες οι οποίοι δείχνουν μία ισορροπία δημοσιονομική και μας επιτρέπουν να προχωρούμε σε αποταμιεύσεις τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούμε βεβαίως και να χρησιμοποιήσουμε υπέρ της ε, οικονομικής ανάπτυξης και της ε, ευημερίας των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε τη σύγκληση συμπληρώνοντας τους θεσμούς μας και το εθεσμικό μας πλαίσιο. Και γι' αυτό είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα εκείνα που θεωρούμε και ξέρουμε ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτήν την ε, οικονομική και νομισματική μας ένωση μαζί με λεπτομερούς τους κανόνες προϋπολογισμού προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό όπως και μια συζήτηση για την επάρκεια του ενωσιακού προϋπολογισμού ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπέρ των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων και υπέρ της σύγκλησης. Με ένα λοιπόν ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο απλώς δεν θα επιτύχουμε πλήρη αποτελέσματα. Είναι σημαντικό όμως να ολοκληρώσουμε αυτό το θεσμικό μας πλαίσιο, αυτούς τους θεσμούς, μεταξύ των άλλων στόχων που σας ανέφερα, προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ κύριος Λούκα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Σεντένο. Σας καλωσορίζω και εξ ε, του ECR. Θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ στην Ελλάδα και στην πιθανή πρόσβασή της ε, στις ε, κεφάλαια αγορές αφού βγει από το τρίτο πρόγραμμα της. Ίσως γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην απόφαση της ε, επί της έκθεσης της ΕΚΤ ζήτησε από την Κεντρική Τράπεζα να περιλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα PSPP αφού έχουν βεβαίως αξιολογηθεί επαρκώς αυτά τα ομόλογα. Χθες όμως είχαμε μία συζήτηση με τον κύριο Τσακαλώτο στην ομάδα δημοσιονομικής βοήθειας όπου τόνισε, βεβαίως ε, αυτό ήταν ένα διαφορετικό ζήτημα μιας προληπτικής γραμμής στήριξης ε, ότι ίσως μια τέτοια προληπτική γραμμή στήριξη ε, είναι το λάθος μήνυμα προς αγορές γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της και δεν εξαρτάται από εξωτερική στήριξη πλέον. Ρώτησα επίσης τον κύριο Τσακαλώτο για την αξιολόγησή του για πιθανές αγορές ομολόγων ε, από την ΕΚΤ μέσω του σχετικού προγράμματος ε, και αν θα ήθελε να πει δημοσίως την ΕΚΤ ότι δεν θέλει η ΕΚΤ ε, να αγοράσει ελληνικά ομόλογα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι εσείς πώς αξιολογείτε το θέμα. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα χρειάζεται και θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις αγορές του, της ΕΚΤ ε, ελληνικών ομολόγων αφού έχει βγει από το πρόγραμμα και πλέον έχουν επαρκή αξιολόγηση τα ελληνικά ομόλογα ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση από την ΕΚΤ να μην περιλάβει στο πρόγραμμα αγορών τα ελληνικά ομόλογα ή θα πρέπει το Eurogroup να κάνει μια τέτοια σύσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Βεβαίω αγοράζουν ε, στη δευτερογενή αγορά. Κλείνει η παρατήση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την ερώτησή σας ε, και για το ότι θίξατε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Το, το θέμα δηλαδή την ανάλυση ε, της κατάστασης της Ελλάδας ε, αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, μπορούμε να δούμε την πορτογαλική εμπειρία. Υπάρχουν δύο βασικές ε, πτυχές εδώ για την επιτυχία αυτών των ε, προγραμμάτων και η Ελλάδα είναι ήδη εδώ και 8 χρόνια σε πρόγραμμα και πρέπει να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που σημαίνει αυτό και την ανάγκη η ελληνική κοινωνία να υιοθετήσει αυτήν την διαδικασία. Το πρώτο λοιπόν είναι πράγματι κάποιοι οικονομικοί όροι και ο μηχανισμός ο ESM και τα θεσμικά όργανα το εξετάζουν αυτό μαζί με τις ελληνικές αρχές και φροντίζουμε στην η Ελλάδα μετά από το πρόγραμμα έχει πλήρη πρόσβαση στις αγορές. Αυτός είναι οπωσδήποτε ο πρώτος όρος, η πρώτη συνθήκη για να επιτύχει η Ελλάδα. Και μετά ε, υπάρχει και μια, ένας εσωτερικός όρος από την πλευρά της Ελλάδας δηλαδή να συνεχίσουν ε, να ε, υπάρχει μια σταθερότητα ανεξαρτήτως ε, του πολιτικού κύκλου για τα ωφέλη του προγράμματος. Συνέβη στην Πορτογαλία, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να αυξηθούν και οι επενδύσεις και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως, η λεπτομερείς διευθετήσεις είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ε, τη στιγμή της εξόδου και οπωσδήποτε εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθούν όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί στην διαδικασία αυτή. Αλλά οι δύο όροι είναι πρόσβαση στις αγορές και ακριβώς ένα κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο είχε και η Πορτογαλία και δημιουργεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό ε, για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και σταθερότητα όπως σας είπα ανεξαρτήτως ε, του πολιτικού κύκλου και πρέπει να το δούμε αυτό ανοιχτά γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικέ και πρέπει να έχουμε όλα τα μέσα στην ερώτησή μας. Μπορείτε να απαντήσετε την ερώτησή μου για τις αγορές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί δεν το απαντήσατε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και η ελληνική κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα. Οπότε, κύριε Λούκη, γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι νομισματική χρηματοδότηση, είναι ένα, είναι ένα μέσο νομισματικής πολιτικής που είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα και την χώρα συγκεκριμένα. Ε, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν ρώτησα εσάς, τον κύριο Σεντένο ρώτησα. Ε, ξεπεράσατε όμως τον χρόνο, είχατε κι άλλο ένα επιπλέον λεπτό. Ε, εν πάση περιπτώσει, κάποια βασικά πράγματα ξεκαθάρισα για να βοηθήσω την συζήτηση να είναι κατανοητή. Και τώρα, κύριος Τρεμόζα. Κύριε Πρόεδρε, καλώ ορίσατε. Προέρχομαι από τους Ελευθέρους. Συγχαρητήρια για την αλέπεια των καθηκόντων σας. Ελπίζουμε ότι θα είναι η συνεργασία μας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τα πήγε πάρα πολύ καλά η Πορτογαλία, η Πορτογαλία που συρρήκνωσε το έλλειμμα Άλλε Άλλες χώρες, ε, Ισπανία και Γαλλία, έχουν πάνω από 3% έλλειμμα την τελευταία δεκαετία. Και αυτό αυξάνεται. Αυτό υπονομεύει την βιωσιμότητα. Ε, αυτό υπονομεύει την πολιτική των επιτοκίων. Εσεί πώς το βλέπετε ως ο νέος πρόεδρο του γύρω Οι κανόνες διάσωσης εφαρμόστηκαν περίεργα γιατί για την Βένετο και για άλλες τράπεζες ε, χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι αλλού. Οπότε Έχουμε τώρα την οδηγία για τις πληρωμές που επίσης έχει εφαρμοστεί διαφοροποιημένα. Και πριν από δύο μήνες εδώ ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Η μη εφαρμογή αυτής της οδηγίας για ε, την υπερημερία που εφαρμόστηκε διαφοροποιημένα. Επίσης για τον Τεγκίντος τι λέτε και την ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως λένε, ε, είχαμε πει εμεί ότι είναι καλό υποψήφιο. Αλλά εμεί πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο το ότι το Eurogroup διάλεξε ένα από τα μέλη του για να πάει να γίνει αντιπρόεδρο της ε, ΕΚΤ. Μα με τέτοια απόφαση τώρα θα έχουμε και άλλους ε, που θα θέλουν μέσω της ΕΚΤ να πάνε στο Eurogroup. Σεντέν. Σας ευχαριστώ κύριε Τρεμόσα για αυτά που ρωτήσατε. Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας είναι ξεκάθαροι. Εφαρμόζουμε το σύμφωνο με ευλάβεια κατά τον ίδιο τρόπο για όλες τις χώρες σήμερα έχουμε όσο γίνεται πιο ομοιογενή κατάσταση από τη μεσογειακή πολιτικής και όσον αφορά τι αποκλήσει των δικτών. Αυτό είναι πολύ καλά μαντάτα για την Ευρώπη. Οπότε η θέση μα είναι αρκετά ισορροπημένη και οι χώρε συγκλίνουν προς αυτό το οποίο έχει εκτιμηθεί ως κατάσταση που συνάδει, συμβαδίζει με τους κανόνες αυτούς και με τους στόχους για όρια ελλείμματος. Ε, σίγουρα πιστεύω ότι και η Γαλλία και η Ισπανία θα βρουν το δρόμο τους σύντομα όσον αφορά αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά Σήμερα έχουμε τους σχετικούς κανονισμούς που είναι αξιόπιστοι, εφαρμόζονται παντού στην Ένωση και αυτά τα οποία αναφέρατε δεν μπορούμε να τα ε, συζητήσουμε τώρα το καθένα, αλλά έτσι ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως το κάθε πρόβλημα ήρθε στη διαφορετική στιγμή όπως και ο κάθε κανονισμός που έχει σχέση με τα προβλήματα ήρθε διαφορετική στιγμή. Φυσικά και περνούν από τη φάση της αναθεώρησης, της τροποποίησης αυτή οι κανονισμοί, έτσι αποκτούν περισσότερη αξιοπιστία, έτσι μειώνουμε τους ε, κινδύνους ε, και επομένως όλα αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει να τα δούμε στο μέλλον όπως και το EPLPS. Είναι ενωπές οι εμπειρίες μας ε, όσον αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση, όσον αφορά την ε, Οικονομική Ένωση, την Νομισματική Ένωση. Θα πρέπει να οριμάσουν όλα αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε εφαρμογή των σχετικών κανόνων με τρόπο ή φόρο που είναι πολύ σημαντικό Τώρα για τον διορισμό του κυρίου Ντεγκίντος στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ συνεχάριν και τους δύο υποψηφίους. Και τους δύο τους γνωρίζω επί πολύ χρόνο και έχω δουλέψει μαζί τους ε, σε διάφορες θέσεις. Σας διαβεβαιώ το βιογραφικό και των δύο υποψηφίων ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ε, εκτιμήθηκε πάρα πολύ από τους υπουργού. Οπότε τελικά η απόφαση διαμορφώθηκε από τα βιογραφικά αυτά. Και θα πρέπει όντως αυτή η δικασία να υπόκειται σε λογοδοσία, να διακρίνεται από διαφάνεια, να, θα πρέπει να μπορούν ε, οι πάντες να μπορούν ανοιχτά να δουν ε, τι γίνεται και να, πώς θα ζυγίζονται ε, τα προσόντα κάθε υποψηφίου. Μίγκελ Βιέγκας. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χτες είχα την ευκαιρία να ακούσω τις παρατηρήσεις σας ε, και απογοητεύτηκα. Μετά από την εμπειρία που είχαμε στην Πορτοκαλία με την Τρόικα όπου είδαμε τα περίεργα αποτελέσματα του Συμφώνου Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης και είδαμε τα όρια ε, που εμπόδιζαν οποιαδήποτε μακροοικονομική σταθεροποίηση τα τελευταία χρόνια και ε, μετά τις αποφάσεις της ε, τελευταίας ε, κυβέρνησης, ακόμα και ενάντια σε αυτά τα οποία έλεγαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θέλω να σας ρωτήσω τι άποψη έχετε κύριε Υπουργέ για τους κανόνες του ευρώ. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις κυκλικές, τις πτυχές αυτών των κανόνων που παρατείνουν ανέτεια την κρίση και τις συνέπειες της. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση που συνδέεται με την πρώτη αφορά ακριβώς το θέμα της σύνδεσης των μελλοντικών προπολογισμών με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Μιλάμε για την δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των ε, συνεπειών ε, των αντικυλικών μέσων που υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τις χώρες ε, που είχαν κολλήσει και πιαστεί στο δίχτυ των κανόνων του ελλείμματος πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι πώς μπορούν οι κυβερνήσεις ε, να προσελκύσουν επενδύσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον και μετά στο θέμα του χρέους οι απαντήσεις που δώσατε χθες ήταν ανεπαρκείς μιλήσατε γενικά αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για τις ιδέες σας για το χρέος. Σας ευχαριστώ. Πράγματι πρέπει να αναλύσει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία πολύ προσεκτικά. Και υπάρχει μια συνεχιζόμενη ανάλυση σχετικά με το πώς λειτουργούν αυτοί οι κανόνες, πώς εφαρμόζονται. Οι κανόνες που ε, συνιστούν δηλαδή το πλαίσιο αυτής της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για την οποία χρειαζόμαστε κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να διέπουν τη στάση των κρατών μελών και τον συντονισμό των οικονομικών εξελίξεων σε όλες τις χώρες. Υπάρχει βεβαίως ένα στοιχείο ευελιξίας στην εφαρμογή των κανόνων αυτών και μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί για το κατά πόσον η ευελιξία αυτή χρησιμοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο αλλά όπως γνωρίζετε το πορτογαλικό παράδειγμα μας δείχνει σαφέστατα ότι είναι δυνατόν να βρει κανείς εναλλακτικές λύσεις εντός του μείγματο πολιτικής όπως το αποκαλούμε που εφαρμόζεται προκειμένου να βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η Ευρώπη δεν έχει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να έχει για να αντιμετωπίζει κρίσεις και οπωσδήποτε δεν τα είχε, ακόμα λιγότερο μάλλον τα είχε, όταν ξέσπασε η κρίση αυτή. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε όλους τους μηχανισμούς να ενισχύσουμε τον μηχανισμό σταθερότητας και αυτό ήταν το βασικό αν θέλετε συμπέρασμα των σχολείων μου και εχθές ότι πρέπει να συντονίσουμε την ανταπόκριση μας, τις απαντήσεις μας, τη διαχείριση κρίσης που είμαστε ικανοί να κινητοποιήσουμε. Η λογική που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να προσπαθούμε με υπομονή να ενισχύουμε τις προσπάθειες των οικοκυριών και των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το δυναμικό τους πλήρως. Και υπογραμμίζω την λέξη υπομονή που είναι όρος κλειδί σε αυτό το πλαίσιο. Μία κρίση χρέους ε, χρειάζεται χρόνια για να την υπερβεί κανείς. και να σας πω ότι η δική μου ερμηνεία του διαλόγου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειαζόμαστε πρόσθετους μηχανισμούς για, τις, για τη χρηματοδότηση και για τις επενδύσεις που να είναι σταθεροί καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου και που να καθιστούν δυνατόν να πραγματοποιούνται στρατηγικά πολύ σημαντικές επενδύσεις στις χρονικές στιγμές που τις χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Σβέν ε, σας καλωσορίζω και εξ ονόματος ε, των Πρασίνων. Η χώρα σας, αλλά και η προσωπική σας ε, συνεισφορά έχει διαψεύσει όσους λένε ότι οι χώρες της ε, Νότιας Ευρώπης δεν μπορούν ε, να ανθίσουν σε ένα κοινό νόμισμα με χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες. Και ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία κάνατε για να κρατήσετε την Ευρώπη Ρωμανική. και διαψεύσατε πολλούς ε, και εντό αυτής της αίθουσας. Παρ' αυτά, ε, σημαντικό είναι το τι θα γίνει όταν θα έχουμε άλλη μια παγκόσμια μακροοικονομική κρίση. Γι' αυτό ζητάμε από σας να είστε φιλόδοξοι στο Eurogroup να ζητήσετε μεταρρυθμίσεις ε, που θα κάνουν ε, το σύστημα ανθεκτικό. Μια που είναι η πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων, νομίζω ότι σημαντικό είναι να μιλήσουμε για τις θεσμικές μας σχέσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα ε, έρχεστε πιο συχνά εδώ από το προκάτοχό σας ε, και αν θα έχετε χρόνο για αυτές τις επαφές με τους ευρωβουλευτές. Δεύτερον, σε μια πρόσφατη σύσταση ο διαμεσολαβητής ε, είπε στο Συμβούλιο ότι υπάρχει κακοδιοίκηση επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια στις θέσεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Τι θα κάνετε για να βελτιώσετε την διαφάνεια στο Συμβούλιο τουλάχιστον εκ των υστέρων για να ξέρουμε τι υποστήριξε το κάθε κράτος μέλος. Η διαφάνεια όταν έχει κάποιος ε, εξουσία έχει μεγάλη σημασία και οπωσδήποτε το Eurogroup ε, έχει μεγάλη εξουσία. Και τέλος ε, κοιτώντα ε, εντό αυτή της ε, θούση ή στο ΔΣ τη ΕΚΤ υπάρχουν λίγες γυναίκες. Τι θα κάνετε για τις επόμενες υποψηφιότητες ε, στην Κεντρική Τράπεζα για να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκίγκολτ, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι σε αυτή τη φάση ακριβώς ε, για τους λόγους που ανέφερα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να έχουμε ε, τιμές απαντήσεις για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Όπως είπα χτες, εγώ θεωρώ ότι οι προκλήσεις για την Ευρώπη ε, θα προέλθουν από το εσωτερικό και το εξωτερικό και οι μεγαλύτερες ε, προκλήσεις ε, και ο κίνδυνος ε, από το εσωτερικό είναι ο κίνδυνος της αδράνειας της χαλάρωσης και της επανάπαυσης πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αυτή τη στιγμή και οπωσδήποτε να τονίσουμε όπως είπατε ε, την πολύ σημαντική αυτή η πολιτική ιδέα των εναλλακτικών. Είναι πολύ σημαντικό σε μια δημοκρατική κοινωνία να παρέχουμε εναλλακτικέ στους πολίτες μας οι οποίες υπάρχουν. Δεν υπάρχει ε, κάποιος μονόδρομος. Πρέπει να τις συζητήσουμε ανοιχτά και τα θεσμικά μας όργανα πρέπει να σχεδιαστούν ε, με έναν τρόπο που να ε, συμμορφώνεται με αυτές τις εναλλακτικές οι οποίες υπάρχουν και ο καλύτερος τρόπος ε, να προωθηθούν αυτές οι εναλλακτικές είναι η διαφάνεια συμφωνώ πλήρως μαζί σας τώρα για την ε, δική μου την διαθεσιμότητα όπως σας είπα και στην αρχή των δηλώσεών μου Σα είπα, είμαι τέλειο ανοιχτός και όποτε είναι αναγκαίο θα μοιραζόμαστε αυτά τα πράγματα μαζί σας. Η διαφάνεια των εργασιών του Eurogroup έχει βελτιωθεί πρόσφατα. Οπωσδήποτε μπορούμε να συνεχίσουμε να την βελτιώνουμε, αλλά βελτιώθηκε πρόσφατα. και κάποιοι εσωτερικοί κανονισμοί που είχαν στόχο να προωθήσουν την διαφάνεια επίσης και ε, οπωσδήποτε θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να είναι σαφής η διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, προστατεύοντάς την βεβαίω, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα αλλά η τα λογοδοσία του που δεν αμφισβητείται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το θέμα των γυναικών. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον καθένα από εμά να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε για τις συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουμε ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ε, υποψηφιότητες όπως ε, η πρόσφατη θέση αντιπροέδρου ε, βεβαίως αξιολογούμε τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αυτό πρέπει να το δούμε στην κάθε χώρα και το κάνουμε αυτό και τώρα μιλώ ως Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας εμείς ε, εφαρμόζουμε έναν κανονισμό ακριβώς για να προωθήσουμε το θέμα αυτό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στην κάθε χώρα Ευχαριστώ Μάρκο Βάλλη Ευχαριστώ Πρόεδρε να καλημερίσω και εγώ τον Πρόεδρο Σεντένο Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς για το μέλλον τη κυβέρνηση τη ΟΝΕ. Ήθελα να ξέρω την άποψή σα ε, για ένα μέσο που θα μπορούσε να ισορροπήσει καλύτερα τα σοκ με αυτό το ποσό που έχουμε πλέον ε, προβλέψει για την απορρόφησή τους εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι μεταφορές, οι δημοσιονομικές, ε, μήπως θα είναι ένα καλύτερο μέσο στο μέλλον αντί για κατά περίπτωση λύσεις που ίσως να μην μπορούν να απορροφήσουν αυτούς τους κραδασμούς στην μια επόμενη δυνητική οικονομική κρίση. Αυτές οι μεταφορές του προϋπολογισμού λοιπόν πώς σας φαίνονται. Για αυτό το European Safe Bond για το οποίο συζητεί η Κομισιόν πλέον, δηλαδή μια τυκλοποίηση του χρέους στην πραγματικότητα, με μια senior και junior επιλογή για τα ομόλογα, δηλαδή junior της ε, περιφέρειας της Ευρωπαϊκής και το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα κουτί της πανδόρας για τις τράπεζες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Περιφέρειας με συνέπειες ε, δύσκολο να που θα ήταν δύσκολο να τις προβλέψει κανείς. Δεν θα ήταν καλύτερα λοιπόν να έχουμε επιτάπητος ένα μέσο που να είναι λιγότερο περίπλοκο και απρόβλεπτο. Επίσης επί των τραπεζών γίνεται μια καλή δουλειά, αλλά δεν βλέπω απτές και συγκεκριμένες ε, πράξεις για τα παράγωγα τα οποία εξακολουθούν να έχουν συστημικές τράπεζες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν στο Eurogroup λοιπόν έχετε κάνει κάτι, έχετε προβλέψει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μελλοντική κρίση αρκετές συστημικές τράπεζες σε σημαντικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Mr. Ευχαριστώ τον κύριο Βάλλη. Δεν θα σας απαντήσω στα Ιταλικά, λέει ο κύριος ε, Σεντένο, για το καλό των συναδέλφων. Είναι σημαντικά αυτά που είπατε. Για το θέμα του προεπολισμού είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε την Ευρωζώνη με κάθε είδους μέσο, όχι μόνο για τη διαχείριση τυχών κρίσεων, αλλά και για τη σύγκληση και για την ενίσχυση των εσωτερικών της κύκλων. Έχουμε συνεργαστεί για να μειώσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε εσωτερικά και πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε και είναι μέρος της δουλειάς που έχουμε μπροστά μας στο άμεσο δηλαδή μέλλον να σκεπτούμε κάποια κονδύλια του προεπολογισμού που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Αυτή η συζήτηση βέβαια θα πρέπει να προχωρεί χέρι με χέρι με τις δυνατότητες χρηματοδότησης του προεπολογισμού και δημιουργίας μονίμων μέσων γιατί αυτός πράγματι είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να προβλέψει κανείς ή μάλλον να κάνει μια προβολή σε μια σταθερότερη αντιμετώπιση και πιο μακροπρόθεσμη. Για το Eurobond αυτό είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο σε επίπεδο κεφαλαίου αγοράς. Ε, όλοι αντιλαμβανόμαστε το πόσο ε, λεπτό είναι το θέμα και πώς αντιδρούν οι αγορές που καμιά φορά αντιδρούν με απρόβλεπτο τρόπο. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν σχεδιάζουμε οποιαδήποτε λύση μπορεί και να χρησιμοποιήσουμε ώστε αυτή η λύση ή αυτό το μέσον να είναι συμπεριληπτικό και να μην οδηγεί σε αποκλεισμό. Και αυτό ισχύει και για τον τραπεζικό τομέα. Προσθέτουμε στον οδικό χάρτη του 16 τα NPL το συζητούμε εσωτερικά υπάρχει μια δέσμη που προετοιμάζει η Κομισιόν προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα κόκκινα δάνεια και είναι σημαντικό αυτό μάλλον και πάλι ένα συμπεριληπτικό και όχι κατακαιρματισμένο πλαίσιο τραπεζικής προσέγγισης είναι σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, λέει ο Πρόεδρος, είχαμε και το EQR και άλλα μέσα. Θα δούμε λοιπόν με ποια συνέπεια θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Για το ο κύριο Μονό. Ολοκληρώσατε την ε, χθεσινή σα εισήγηση γιατί ποτέ χρειάζεται περισσότερο δημοκρατικός έλεγχος στην ΩΝΕ. Αυτό ε, ελπίζουμε να μην ευσεβείς πόθος. Από το 1992 δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από τον κόσμο επί της ΩΝΕ. Έχω τρεις έρευνες. Η κεντρική τράπεζα μέσω του ΣΣΜ πρόκειται να δημιουργήσει κάποιες πρακτικές πάρα πολύ αμφίβολες και έτσι επομένως θα υπάρξει ένα πρόβλημα για τις μικροεπιχειρήσεις όσον αφορά τον δανεισμό τώρα που τα έχουν βρει δύσκολα. Επίσης η σχέση μεταξύ των τοπικών οικοσυστημάτων και των τραπεζών ε, έχει δυσκολέψει και με το SSM πρόκειται να χάσουν αυτές οι περιοχές 0,2% του ΑΕΠ και η νομική υπηρεσία έχει πει ότι ο SSM ε, ε, ε, κατησχεί και παρακάμπτει την νομοθεσία. Πρόκειται να υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες στο Κοινοβουλίο αλλά μέχρι τώρα το έχει αγνοήσει ο SSM το Κοινοβουλίο. Για πέστε μας εσείς ε, πώς τα βλέπετε. Δεύτερον, όσον αφορά την Λετωνία, με κάθε επιφύλαξη για τις νομικές ε, εξελίξεις, η κοινή γνώμη λέει ότι κανένα πολιτικός δεν μπορεί να υποχρεώσει σε παρέτηση κάποιον κεντρικό τραπεζίτη. Πρεσμένη εβδομάδα όμως το Eurogroup ε, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά αυτό φύγει όλη την Ευρώπη. Μια που ο άνθρωπος αυτός ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Μα τι γίνεται, δεν υπάρχει ούτε στην Κεντρική Τράπεζα Δημοκρατικός Έλεγχος. Τέλος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το περίφημο νομισματικό ταμείο όσον αφορά τους νέους φορείς που επίσης ε, εκφεύγουν παντός ελέγχου ως πρόεδρος του Eurogroup για αυτό το νομισματικό ταμείο τι δημοκρατικό έλεγχο θα προβλέψετε. Σεντένο. Ευχαριστώ κύριε Μονό. Αυτά που είπατε σχετίζονται με κάτι σημαντικό όσον αφορά την θεσμική αρχιτεκτονική και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα κάνουμε. Προς κάθε κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει προσοχή. Όσο αφορά την εξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, έχω να σας πω ότι καταλήξαν σε τέτοια ρακεκτονική θεσμική ούτως ώστε για την νομισματική πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει ανεξαρτησία. Σε τέτοιο βαθμό όλα αυτά να συνάδουν με τη σιγουριά που θέλουμε να έχουμε όσον αφορά την χρήση των μέσων πολιτικής που διαθέτουμε. Άρα θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει αυτή η ανεξαρτησία ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η αξιοπιστία για την πολιτική μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υποχρέωση λογοδοσία για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το μέτωπο. Ναι, είναι σημαντικά αυτά τα οποία είπατε και θα τα λάβουμε υπόψη. Και όσον αφορά τι αποφάσει για την χάραξη τη πολιτική, ακριβώ είναι σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία. Τώρα τον προπολογισμό και το EMF. Συζητείτε τώρα το θέμα. Συζητήσεις είναι σε εξέλιξη. δεν θα σταματήσει η δημοσιομική εποπτεία. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ορίζει ξεκάθαρα τι ισχύει. Και ούτε θα πρέπει να υπάρχει για το ΕΜΕΦ ή ΕΣΕΜ κάποιο είδου επικάλυψη μετά του Συμφώνου σταθερότητα. Μιλάει ταυτόχρονα ο πρόεδρος με τον κύριο Μονό. Συμπαθάτε με γιατί δεν έχουμε χρόνο, οπότε ε, τώρα έκλεισε ο πρώτος κύκλος των ε, αγορεύσεων της πολιτικής ομάδας και τώρα πάμε στο δεύτερο κύκλο τέσσερα λεπτά έκαστος και θα δώσουμε τώρα το λόγο σε όλους τους Σαν που θέλουν το λόγο, αν Σαντέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε και εσείς Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων την τόσο ενδιαφέρουσα για σήμερα το πρωί. Είπατε τι γίνεται με τους μεγαλογονομικούς δείκτες που έχουν απογειωθεί, είναι στο πράσινο, κάτι το οποίο πολύ θετικό και έχουμε ρυθμό ανάπτυξης για το 2,5% ε, και έχουμε ελλείμματα τα οποία συρρυκνώνονται ακριβώς όπως και η ανεργία. Έχουμε δε τις ε, μεταρρυθμίσεις που προχωρούν, ε, επίση την διθάσευση των ε, δημοσίων δαπανών, άρα πολύ καλές επίδοσεις. Θα πρέπει τα κρατημέλη να μειώσουν τα ελλείμματα, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο χρέος το οποίο ε, είναι το ευκταίο. Και αυτά σας τα λέω με τα λόγω γιατί αυτό είναι πρόβλημα της δικής μου χώρας. Τώρα όσον αφορά την αποπληρωμή των σχετικών χρεών αυτό είναι σημαντικό ε, ούτως ώστε να έχουμε επενδύσεις, να έχουμε ανάπτυξη και επίσης ε, έχουμε τώρα χαμηλά επιτόκια Εάν τα επιτόκια αυξηθούν, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Το Eurogroup βεβαίως και επεξεργάζεται όλα αυτά τα θέματα, γνωρίζετε το θέμα ή τα θέματα και για πέστε μας τι μπορείτε να κάνετε, ε, πώς μπορείτε να βοηθήσετε, πώς, πώς θα κάνετε προτεραιότητα τη συρρήκνωση του χρέους, πώς θα εξοηθούν τα κρατημέλη να λάβουν τα πιο σωστά μέτρα, γιατί το έχουμε συζητήσει Τότε χρειάζεται τα κράτη-μέλη με υπευθυνότητα να κάνουν τέτοιες προσπάθειες, να είναι και αλληλέγγυα. Έχουν τη σχετική ευθύνη τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Σύνδερο, σας ευχαριστώ κυρία Σαντέ. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτό ακριβώ που είπατε. Τι σημασία του πώς θα εξυπηρετηθεί το χρέος. Γιατί περνάμε τώρα μια μαθηματική περίοδο και είναι αλήθεια ότι οι οικονομικοί δείκτες γενικώ πάνε καλά. Δημιουργήθηκαν τώρα πρόσφατα πάνω από 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και πώς απλά το χρέος ας κατανοηθεί ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες ασυμμετρίες στην Ευρωζώνη. Αλλά είναι σημαντικό όλες οι χώρες και κάθε μία χωριστά να αρχίσουν να μειώνουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Η κρίση είχε πολλές συνέπειες επηρεάζουν και το μέλλον και από ό,τι γνωρίζουμε από παλιότερες κρίσεις ε, το πιο σημαντική στιγμή είναι όταν αρχίσει αυτός ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να συρρυκνώνεται και άρα το πιο σημαντικό είναι έτσι να βοηθήσει κανείς την ανάπτυξη και έτσι να εξασφαλίσουμε το ότι όλες οι χώρες θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε μια ματιά στα στοιχεία για τις πρόσφατες εξελίξεις. Θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότερες χώρες ήδη έχουν πάρει αυτή την κατεύθυνση. Είναι σε αυτή τη φάση και έχουν τέ, τέτοιου είδους κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος Πολ Τάνκ. Ευχαριστώ κύριε Σεντένο που ήρθατε και συγχαρητήρια γενικότερη ερώτηση. Τι μάθατε από τον προκάτοχό σας, τον κύριο Ντάσσελμπλουμ. Εντάξει, συνένωσε την ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να οικοδομήσει πιστοσύνη. μεταξύ Βορρά και Νότου. Θυμάμαι κάτι παρατηρήσεις του για γυναίκες και ποτά και την κατακραυγή που δημιούργησε και οπωσδήποτε είναι ένα καλό σημάδι. Και βεβαίως ε, ζητήματα όπως η Τραπεζική Ένωση, η Δημοσιονομική Ικανότητα της Ένωσης που απαιτούν εμπιστοσύνη μεταξύ Βορρά και Νότου. Ε, τι θα κάνετε λοιπόν για να γεφυρώσετε αυτό το κενό. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με την ε, διαφάνεια. Έχουμε εδώ μια περίπτωση που αφορά και διορισμό στο ΔΣ της ΕΚΤ ε, ότι συζητήθηκε στο Eurogroup αλλά θα τοποθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι θα κάνουμε λοιπόν με την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι και μέρος της δημοκρατικής διαφάνειας ε, να έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Τάγκ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι δύσκολη δουλειά. Και οπωσδήποτε σκοπεύω να πάω προς μια συνενετική κατεύθυνση στο Eurogroup και αυτό είναι το πιο σημαντικό θα έλεγα πολιτικό ζήτημα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας πω ότι θεωρώ ότι καμιά φορά εμείς οι πολιτικοί μεγενθύνουμε τις διαφορές μεταξύ Βόρα και Νότου για τους δικούς μας ε, σκοπούς ε, και τις διωγγώνουμε. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, το ανέφερα αυτό πολλές φορές ήδη έχουμε οικοδομήσει την Ευρώπη ως ένα πολιτικό εγχείρημα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης αυτό ε, χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση έχουμε τώρα την δυνατότητα να αξιολογήσουμε το πόσο σημαντικές είναι οι κοινέ μας αποφάσεις ε, προς όφελος των πολιτών μας γιατί αντιμετωπίσαμε μια πολύ δύσκολη κρίση και καταφέραμε να επεκτείνουμε το θεσμικό πλαίσιο και να έχουμε την επιτυχία που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση είναι ε, πολύ ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα αυτά στις χώρες μας το αντιλαμβάνομαι πρέπει να καθορίσουμε θα έλεγα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και εντό αυτού να βρούμε λύσεις ε, που μας ε, ικανοποιούν και βεβαίως έχουμε τον ε, γενικότερο στόχο να αυξηθεί δηλαδή η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης και όλοι ωφελούμαστε από αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε ότι έτσι θα ε, γίνεται και στο μέλλον για την ε, διαφάνεια το ανέφερα και πριν σε σχέση με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ ακολουθήσαμε τον κανονισμό ο οποίος ε, μιλάει για επίσημη ακρόαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα λάβει χώρα ε, προσεχώς είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις ε, εκ των προτέρων και με τους υποψηφίους αυτό προβλέπει ο κανονισμός οπότε νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ε, πάντα βεβαίω με πολύ βάθο εξέταση αυτά προβλέπω κανονισμό αυτή τη στιγμή ευχαριστώ Ότμαρ Κάρα. Κύριε Πρόεδρε συγχαρητήρια για τον διορισμό σας ερώτηση μου είναι εξή. Αυτή τη στιγμή είμαι σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ για το πακέτο μείωση του κινδύνου και κάποιοι θεωρούν ότι ένα ξεκάθαρο κατόφλι θα πρέπει να καθοριστεί ειδικά όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πριν γίνει ο μηχανισμός επιχειρησιακός. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό ε, δεδομένων και των αποτελεσμάτων της πρώτης έκθεσης προόδου ε, για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Κομισιόν τον Ιανουάριο. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ποιο όραμα έχετε για να αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Για την ερώτησή σας ευχαριστώ. Ο δικός χάρτης 2016 ορίζει τις περιοχές στις οποίες να κινηθούμε προς τα εμπρός για τη μείωση του κινδύνου. Υπάρχουν αρκετές δέσμες που ήδη υπευλήθησαν από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκαν και νομίζω ότι θα εκπληρωθούν τα κριτήρια της μείωσης του κινδύνου ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και στα υπόλοιπα μέτρα μετρίασης του κινδύνου. Αυτό θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από μία μόνιμη αξιολόγηση του προόδου που σημειώνεται στη μείωση του κινδύνου για τη μείωση και τη συγκράτηση των NPL όπως ανέφερα και εγώ και ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη για την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών 460 δις ευρώ εδόθησαν από την αρχή της κρίσης της τράπεζης. και η μείωση του κινδύνου και η στήριξη και των ιδιωτικών και των ε, δημοσίων φορέων στην Ευρώπη υπήρξε από την αρχή ε, προτεραιότητα και κάτι που πρέπει και μπορεί να δώσει ε, περισσότερη εμπιστοσύνη για τον μηχανισμό σταθερότητας συζητούμε το πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη λειτουργία του προκειμένου να τον πρικήσουμε με περισσότερα μέσα διαχείρισης κινδύνου ώστε να είναι πιο ανθεκτικός στο μέλλον. Το θέμα που αναφέρατε έχει σχέση με την ανάπτυξη, με την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό όλα τα μέλη της Ευρωζώνης να αισθάνονται άνετα καλυμμένοι από τη λειτουργία αυτών των θεσμών. Δεν μιλούμε για έλλειψη λογοδοσίας βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Η προσωπική μου επιλογή, για να σας το πω ειλικρινώς, θα ήταν πρώτα να συζητηθεί η ουσία και μετά αυτό που λέτε. Και βεβαίως ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα υποστηρίξουν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη αυτού του εργαλείου ή στον προϋπολογισμό Ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα χρειαστείτε κύριε Σεντένο τα ακουστικά σας εκτός αν ξέρετε ελληνικά. Σήμερα είναι και η, η, μέρα της μητρικής γλώσσας. Θα σας συγχαρώ, γιατί στα στο αρχικό σας statement έχω κρατήσει τρία πράγματα. Democratic accountability, πάρα πολύ σημαντικό. growth that is inclusive δεν υπάρχει λόγος να το εξηγήσω. Και το τρίτο, deepening of the EMU with completion of the banking union. Εγώ θα σας ρωτήσω δύο ερωτήματα, πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί τέθηκαν από συναδέλφους μου, αλλά σε πιο γενικό επίπεδο. Από το Γενάρη του 2013, που τέθηκε σε ισχύ το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, μέχρι σήμερα το αποτέλεσμα σε επίπεδο πραγμα... σύγκλησης της, της πραγματικής οικονομίας είναι απογοητευτικό. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Το πρώτο μου ερώτημα είναι ότι ενώ δόθηκε μεγάλη φροντίδα, μεγάλη προσοχή στα ελλείμματα των κρατών μελών, δεν δόθηκε σημασία στα πλεονάσματα, που είναι μέρος του προβλήματος. Μάλιστα κάποιοι έχουν και την άποψη ότι εν πολλής τα ελλείμματα είναι και αποτέλεσμα των πλεονασμάτων. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Και το δεύτερο είναι σχετικά με τα NPLs. Έχει ήδη τεθεί το θέμα και εδώ όμως θα είμαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Αναγνωρίζουμε οι περισσότεροι εδώ ότι τα NPLs δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τις τράπεζες, μας αφορά όλους, σαν Ευρωζώνη, σαν θεσμούς της Ευρωζώνης. Είστε υπέρ, ε, τίθεστε ευνοϊκά στη δημιουργία uh, bad banks, αυτού του asset management tool. Αυτό θα ήθελα να γνωρίζω, γιατί αφορά πάρα πολλές κράτη και τραπεζικά συστήματα στην Ευρωζώνη. Σας ευχαριστώ και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας. Και θα είμαστε δίπλα σας επικοδομητικά κριτικά. Oh, Ευχαριστώ τον κύριο Μαυρίδη για την ε, ερώτηση και την παρατήρηση και για τον τρόπο με τον οποίο ε, αξιολογείτε εσείς τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. η σύγκληση που έχουμε παρατηρήσει και η ονομαστική και η πραγματική γιατί αντιμετωπίσαμε πολύ ουσιαστική κρίση σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιολογείται δηλαδή η κρίση κατέστησε πολύ πιο δύσκολη όλη αυτή την προσπάθεια σύγκλησης ακόμα δε περισσότερο όταν όπως ήδη ανέφερα έχουμε αυτό το αν μη πλήρες εν περιπτώσει θεσμικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει στη σύγκληση να λάβει χώρα να υλοποιηθεί με πλήρη τρόπο στα πλαίσια μιας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Οι διαδικασίε λοιπόν είναι πολύ βραδίες, η υπομονή που ανέφερα νωρίτερα είναι πάρα πολύ σημαντική από όλους και για όλους αλλά πρέπει να υποστηρίζουμε όπως μπορούμε τη σύγκληση. Στην διαδικασία μακροοικονομικών ε, ε, ασταθειών και στην περίπτωση των πλεονασμάτων και στην περίπτωση των ελλημάτων και κοιτώντας την περιοχή στο σύνολό της, κοιτώντας δηλαδή τις εξωτερικές, τα εξωτερικά σημεία αστάθειας, πρέπει να βλέπει κανείς το άθροισμα του πλεονάσματος μαζί με τις εξοικονομήσεις που θα πρέπει να επενδύονται στην Ευρωζώνη και να ε, καταλήγουν σε όφελος για όλα τα μέλη. Τώρα μας πιέζει και ο χρόνος όπως βλέπω. Τα NPL, τα κόκκινα δάνεια, πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκουν στην πραγματική οικονομία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν πώς θα αντιμετωπίζουμε ώστε να διατηρούν, να διατηρείται η πραγματική αξία της ε, οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν κάθε χώρα να αντιμετωπίζει με μεγάλη προσοχή και σύμφωνα με το δικό της πλαίσιο και τις δικές της δυνατότητες τα στοιχεία αυτά. Γιατί κάποια από αυτά, τα μη εξυπηρετούμενα, εν πάση περιπτώσει, δάνεια, έχουν πραγματική οικονομική αξία. Είναι όμως μια ευρεία συζήτηση. Πρέπει να δουλέψουμε εντός των κανονισμών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα του BRID, αλλά μια συζήτηση που θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύμφωνα με τα προγνωστικά της Κομισιόν του 2018, η πρωτοβουλία θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης κάτω του μέσου όρου. Απόκληση επομένω. Και άλλα κράτη-μέλη που ήταν σε παρόμοια κατάσταση όπως η Ιρλανδία πρόκειται να έχουν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από όσο η Πορτογαλία. Και η Ελλάδα. Και εκεί προσέχει ταχύτητα του ρυθμού ανάπτυξη. Και σα ερωτώ, ως πρόεδρος του Eurogroup τι θα συνιστούσατε στον Υπουργό Οικονομικών της Πορτογαλίας για να ανατρέψει αυτή την τάση. Σέντερ, ευχαριστώ. Κύριε Φερνάντες, ως πρόεδρος του Eurogroup αυτό το οποίο εγώ θα συνιστούσα σε όλους τους οικονομικών της, Euro, της Ευρωζώνης να συνεχίσουν την προσπάθεια που ήδη έχουν ξεκινήσει. Να συνεχίσουν να επιδιώκουν την σταθερότητα όσον αφορά τα οικονομικά, σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα και να προσπαθούν να βοηθήσουν στην ανταγωνιστικότητα του συνόλου της Ευρωζώνης. Σήμερα Βρισκόμαστε σε μία περίοδο ανάπτυξης που είναι ρεκόρ, θετικό. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και για την Πορτογαλία. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια διάρκεια ανάπτυξης και άρχισε η Πορτογαλία το 2017 να συγκλίνει προς τον μέσο της Ευρωζώνης. Για να δούμε πώς θα πάμε το 18. Πάντως, εγώ θα πολύ ικανοποιημένο εάν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης ήταν στη θέση να εκπληρώσουν τις ε, προβλέψεις μας. Ναι, ναι, ναι, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο, στο μέσο όρο του ρυθμού ανάπτυξη. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Γκουαλτιέρ, και το λόγο στον κύριο Χώνα Φεράντε. Ευχαριστώ, πρώτο, ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την ανάπτυξη καθηγόντων σας και επίσης μπράβο για το έργο σας ε, στην ε, Πορτογαλία γιατί πέραν του, του καλού που κάνατε στους συμπατριώτες σας δώσατε ελπίδες σε όλη την Ευρώπη. Και επανειλημμένα έχετε πει ότι θέλετε να συνδυαστεί η φιλοδοξία με την ε, υπομονή και αυτός ο συνδυασμός πολλές φορές όμως δεν είναι εφικτός για μας σε σχέση με διάφορα νομοθετήματα όπως το έντις για την ασφαλεία των καταθέσεων. Έχει πράσει μια διαδικασία συνομιλιών με το Συμβούλιο και ο συνέδρος Μπάλτς ε, λέει και ξαναλέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα πακέτα συρρήγνωσης των κινδύνων και εγώ δεν έχω αντίρρηση αυτό που είπε αλλά αυτές τις μέτρων τελικά παρελκύουν τη συζήτηση και στο Συμβούλιο και εδώ και επομένως Πάμε πολύ αργά. Εντάξει, είναι θέμα του ΕΚΟΦΗΝ, αλλά για να μας εσείς ως πρόεδρος του Γιώργου. θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο τόσο ώστε να πιέσουμε, τόσο ώστε να μπορέσουμε να, να τα πράγματα, να, να υπάρξει αυτός ο εγωνισμός και να μπορέσουν ε, ε, οι μεν και οι δε να τα βρουν ε, για να μπορέσει να μας βοηθήσει ε, αυτός ο συνδυασμός ε, φιλοδοξίας και υπομονής. Εμείς είμαστε ανυπόμονοι για αυτόν τον κανονισμό. Τι να κάνουμε για να σπρώξουμε λίγο τα πράγματα. Σεντένα. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Ναι, όντως χρειάζεται να υπάρξει η υπομονή. Γενικά να διαπνέει υπομονή το σύστημα. Παρακαλώ να αντέξετε λίγο παραπάνω. Αλλά καμιά φορά ναι, και η ανυπομονησία δίνει όθηση στα πράγματα και βοηθά στην λήψη αποφάσεων. Αυτά. Τελικά. Γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Κατάλληλη οικονομική και πολιτική συγκυρία. Δηλαδή να προωθούν αυτοί οι κανονισμοί, ε, αυτές όλες οι προτάσεις να έχουν αίσια κατάληξη για να ακολουθήσουμε αυτόν τον δικό χάρτη. Συμφωνώ μαζί σας. Ε, ώρα ήτανε, ούτως ώστε να κινηθούν τα πράγματα ως πρόεδρο του Eurogroup. Όσο μπορώ. Θα συμβάλλω στο να προχωρήσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Να μπορέσουμε τον Ιούνιο να προσπάσουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτό το μέτωπο. Ο Γκολτιέρη, κάτσε διάει δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ένα λεπτό καθένας κύριε Παπαδημούλη. Κύριε Σεντένο, σημείωσαμε ιδιαίτερη ικανοποίηση Κύριε Σεντένο, σημείωσαμε ιδιαίτερη ικανοποίηση τα εξαιρετικά θετικά σχόλια που κάνατε για τη χώρα μου την Ελλάδα, τις ελπιδοφόρες εξελίξεις που μας ανακοινώσατε και κράτησα και τη δήλωσή σας μετά το Eurogroup προχθές που είπατε τώρα η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο. Επειδή έχετε θέσει ένα πολύ φιλόδοξο και πυκνό χρονοδιάγραμμα η ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει τη δική της στρατηγική ανάπτυξη με τις μεταρρυθμίσεις και τα υγιή δημόσια οικονομικά για μετά το τέλος των μνημονίων, τον Απρίλιο, και εσείς να εξειδικεύσετε τα μέτρα ελάφρυσης του χρέους που έχετε αποφασίσει από τον Ιούνιο, μέσα στον Απρίλιο, να ολοκληρώσετε και την τέταρτη αξιολόγηση και όλα αυτά να έχουν τελειώσει τον Ιούνιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μας παρουσίασε χθε ως συμφωνημένο στο Eurogroup ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα από πλευράς δική σας και τι σημαίνει η μπάλα στο δικό σας γήπεδο, τι σκοπεύετε να κάνετε για να τελειώνουμε με αυτή την περιπέτεια. Ε, θα ήθελα να παραμείνω και θα είμαι πάντα θετικός ε, για τις ε, εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα. Βλέπουμε πολύ αποφασιστική και παραγωγική δουλειά από τις ελληνικές αρχές για την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως είπα στην εισαγωγή μου η έκφραση ότι τώρα η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο αφορά διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν ε, από τις ε, χώρες για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση όσον αφορά την εκταμίευση και γι' αυτό ακριβώς ε, παρακινούσα και τις χώρες να κινητοποιηθούν και οι αντιδράσεις που είχαμε στο Eurogroup ήταν πολύ θετικές ως προς αυτό οπότε δεν έχω κάποια αμφιβολία ότι θα επιτύχουμε στην ολοκλήρωση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νίνα Γκίλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ε, συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου. Ε, κάτι θα ήθελα να πω γρήγορα. Ε, η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται και ο ήλιος λάμπει αλλά αν το δούμε αυξάνεται και η ανισότητα στην Ευρώπη 40% του πλούτου βρίσκεται στα χέρια του 1% και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό ένα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογέ ε, πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα 120 εκατομμύρια άνθρωπους που είναι φτωχοί 20 εκατομμύρια παιδιά που είναι κατά το όριο της φτώχειας ε, θεωρώ λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια ευκαιρία για την ε, Κομισιόν ε, να έχει μια στρατηγική μείωση της ανισότητας. Πώς θα προσπαθήσετε λοιπόν να έχετε κάποιες μεταρρυθμίσεις ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, λίγο Πρόεδρος. Ε, τοποθετηθήκατε με συντομία σε ένα ευρύτατο ζήτημα. Σα ευχαριστώ που το θέτετε. Είναι σημαντικό να προωθούμε στρατηγικές ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνουν τους πάντες. Αντιμετωπίσαμε υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, το οποίο ήταν καταστροφικό, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις οικονομίες μας ήταν και πηγή ένδυας. Επομένως, χρειαζόμαστε δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες των αγορών μας απασχόλησης, ιδιαίτερα ως προς την νεολαία, για να δώσουμε προσδοκία στις αγορές μας και στις χώρες. Υπάρχουν ανισότητες, χρειάζονται μέτρα, μέτρα σύγκλησης και επομένως η προηγούμενη συζήτηση για την πρόθεση της σύγκλησης εντός της Ευρωζώνης είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είναι σημαντική και καθοριστική και για το μείγμα πολιτικής μας. Θα εξετάζουμε λοιπόν οπωσδήποτε τα θέματα υπό αυτήν την οπτική της συμπεριληπτικότητας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σεντένο βεβαίω για αυτό το θαυμάσιο ξεκίνημα του διαλόγου και της συνεργασίας μας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυναντηθούμε σύντομα και να ανακοινώσουμε και τις μεθόδους εργασίας μας ώστε να έμπρακτα μάλλον να υπογραμμίσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη επιφάνεια και διαφάνεια όμως σε αυτόν τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της οικονομικής μας πολιτικής. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε αν θέλετε γιατί έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε τώρα τον, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών και την Ετήσια Επισκόπηση. Θα ψηφίσουμε το απόγευμα. Έχουμε τον, κύριο, τον εισηγητή, τον κύριο Μπαγιέ, και θα ξεκινήσω δίνοντας του 5 λεπτά για μια εισαγωγική τοποθέτηση. Ε, Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον νέο Πρόεδρο. Καταρχά ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που με επέτρεψαν να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ήταν μια δύσκολη θεματική εξέταση πολύ συχνά οι πολιτικέ ομάδες είναι πολύ απομακρυσμένε Εδώ νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα καλό συμβαστικό κείμενο. Και νομίζω ότι αυτό το κείμενο που θα ψηφίσουμε το απόγευμα είναι μια πραγματική πρόοδος γιατί μας δίνει απτές λύσεις για να μειώσουμε τις ε, κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες να περιορίσουμε την ένδυα των εργαζομένων και να αυξήσουμε τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αυτή η μεγέθυνση αρχίζει να γίνεται πιο αισθητή. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης απασχόληση βεβαίως και έχουμε ακόμα δυναμικό ε, μεγέθυνσης που πρέπει να το αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα ενεργειακά αλλά βεβαίω οι κοινωνικοί, και οι οικονομικοί στόχοι τη απασχόληση παραμένουν οι πιο σημαντικοί. Πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε στις διάφορες ε, ταχύτατε εξελίξεις τη διεθνού αγορά, Πολύ συχνά οι εργαζόμενοι είναι τα πρώτα θύματα του αυτών των ε, διακυμάνσεων. Ξεκινώ λοιπόν με μια ανάγκη αύξησης των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων που θα πρέπει να κατευθύνονται στην προγραμματική οικονομία γιατί γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις είναι αρκετά περιορισμένες. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα εμπόδια για την υλοποίηση μεγάλων έργων επενδυτικών και την πρόθεση εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού δημοσίου δικαίου, το οποίο βέβαια καμιά φορά αντιμετωπίζει και τα δικά του προβλήματα. Στις υποδομές όμως και στην υγεία ιδιαίτερα δεν έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις και αυτό οδηγεί στην δημιουργία θέσης, θέσεων απασχόλησης. Επίσης χρειαζόμαστε υπεύθυνε επενδύσεις σε τα δημοσιονομικά και στην Ευρωζώνη θα πρέπει να οδηγούν σε βιωσιμότητα και καλή διαχείριση. Υπάρχει και η πρόταση της αύξησης ε, της μισθολογικής ε, που έχει υποστηριχθεί και από τον πρόεδρο Ντράγκη για να επανεκκινήσουμε στο σύνολο της νευρακή οικονομία εκπαραλλήλουμε μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το παρελθόν ε, για την ελάφρυνση του άχθους. Χρειάζονται και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίσουμε και το εγγυητικό μέσο για τους νέους, ε, ε, την πολιτική για τις επιχειρήσεις, για την παιδεία και για την κοινωνική ασφάλεια. Στην ουσία όλα αυτά που συνιστούν την προσθέμενη αξία της δικής μας υπήρου έναντι των υπόλοιπων περιοχών του κόσμου. Πρέπει να την προστατεύσουμε αλλά και να την βελτιώσουμε αυτήν την προσθεμένη αξία για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνώνυμο ελπίδας. Μιλούμε και για τον ε, δημοσιονομικό ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το φορολογικό μάλλον ανταγωνισμό που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και ομίλους να επιλέγουν που θα εγκαθίστανται. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και θα πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα πιο κοινό φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. Και στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης ε, εξετάζουμε την ε, καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων φορέων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και των ε, θεσμικών αλλά και των εταίρων και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων φορέων που θα μας επέτρεπε μια καλύτερη εφαρμογή των ε, αναχώραση τάσεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια θετική ψήφο σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή μας. Περνάμε τώρα στους ομιλητές. Ε, τρία λεπτά ο καθένας. Τόμ Φάντερ Καντελάρε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Ιγ Μπαγιέ για την ε, φοβερή δουλειά που έκανε. Χρειάστηκε βεβαίω ε, λίγο χρόνο για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, αλλά τελικά είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε συμβαστικέ προτάσει που θα υποστηριχθούν, ελπίζω, στην ψηφοφορία το απόγευμα. Και θα ήθελα να τονίσω ε, τι άπνε προσπάθειε του Ιγκμπαγιέ και των λοιπόν ε, συναδέλφων. Επίση, το ΕΛΚ θα υποστηρίξει όλε τι συμβαστικέ προτάσει και στην τελική έκθεση και από πλευράς δομή ε, και περιεχομένου έχουν ληφθεί υπόψη κάποια πράγματα. Θα ήθελα να τονίσω τρία από αυτά. Πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις υποβάλαμε ως Κοινοβούλιο ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Μια ισορροπία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ψηλότερε επενδύσεις ε, θα οδηγήσουν σε αύξηση τη ζήτηση ε, και επίση τονίζουμε την σημασία του να αποφευθούν οι στενοποί επενδύσεων, ειδικά στο Βέλγιο τα βλέπουμε κάθε μέρα αυτά, όταν έχουμε κολλήσει στο μποτιλιάρισμα. Το δεύτερο ζήτημα που ανέφερα αφορά ακριβώς ε, τα θέματα της δημόσιας χρηματοδότησης. Όπως ξέρουμε δεν υπάρχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Ε, πιο συγκεκριμένα νομίζω ότι οι παρατηρήσεις για τους πληθυσμούς που γυράσκουν ε, και για τα κράτη-μέλη που πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους ε, νομίζω είναι πολύ σημαντικά μηνύματα που περιέχονται στην έκθεση. Τρίτο και τελευταίο. Χαίρομαι που τονίζονται και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές προσελκύουν επενδύσεις και αυξάνουν τα πραγματικά εισοδήματα και βεβαίως τονίζεται και το ζήτημα των αγορών εργασίας και του μέλλοντος της εργασίας και εδώ πέρα πραγματικά πτυχαίνουμε μια ισορροπημένη αλλά και ουσιαστική ε, άποψη και βέβαιως έχουμε και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, ε, δύο λόγια για το μήνυμα μας ε, για την στάση της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι είναι θετικό το ότι κάνουμε αναφορά και στην ε, στάση της Ευρωζώνης. Ε, και συνολικά χαίρομαι για το μήνυμα που στέλνει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά που έκαναν. Ευχαριστώ Τόμ ευχαριστώ και για τις ε, πληροφορίες αυτές. Παίρναμε τώρα στο ECR. Μπέρντ Λούκε, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, Ιγκμπαγέ για την συνεργασία που είχαμε. Πράγματι αρχικά η έκθεση ε, μας είχε φανεί ως μια έκθεση με την οποία δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αλλά τελικά είχαμε πάρα πολύ θετικές συζητήσεις και πολύ θετικό πνεύμα του εισηγητή Συνολικά λοιπόν θα έχουμε πολύ καλές ε, συμβαστικές προτάσεις με τις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε Και βεβαίως χαιρόμαστε ε, το ότι τονίζεται εδώ πέρα το πλαίσιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου, του πλέγματος ευθύνης ε, και ανάληψης ε, των συνεπειών και βεβαίως γίνεται νομίζω και μια αναφορά στις ανισότητες, στην εξέλιξη της Ευρωζώνης. Ε, έχουμε βρει εδώ πέρα λοιπόν πάρα πολύ ε, σωστές ε, διατυπώσεις ειδικά όσον αφορά τις στοχότερες χώρες της Ευρωζώνης ταυτόχρονα η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και ανισότητας δεν αναφέρεται επαρκώς και νομίζω ότι έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και νομίζω ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις οι οποίες μπορέσαμε να, συμφων... να συμβιβάσουμε τελικά γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ευχαριστώ Thank you very much and also... Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον ε, εισηγητή που έδειξε τέτοιο πνεύμα συνεργασίας Α, βλέπω αντί του αντί της Καρολίνα είναι εδώ ο κύριος Τρεμόσα. Δεν μπορεί να είναι εδώ η Καρολίνα, αλλά είπε ε, σε μένα να πω ότι ευχαριστώ όλους τους και οδησυχητές και τον εισηγητή για την συνεργασία των τελευταίων εβδομάδων. Επίσης, υπενθυμίζει ότι η Άλντε στηρίζει τους περισσότερους συμβασμούς και βέβαια θέλαμε εμεί ω ομάδα να τονιστούν οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι τουλάχιστον μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα κείμενο πιο ε, ισορροπημένο στι τελευταίε εβδομάδε. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα, ή θα πρέπει να είναι δεσμευτικές ή δεν έχουν νόημα. Γιατί τα κρατημέλη τις αγνοούν. Το είδαμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν πιάνει τόπο καμία σύσταση. Άρα, ή δεσμευτικέ ή αχρίαστες. Κάθε χρόνο τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για την ΚΟΕ. ουρμπαν Ούρμπαν Κρέσπο. Έχετε τρία λεπτά. Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πούμε μπράβο για την προσπάθειά του στον εισηγητή. Προσπάθησε να φτιάξει κείμενο το οποίο να καλύψει όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, έχει αυτή την ε, κριτική άποψη για το τι έγινε αυτό το εξάμεινο, τι γίνεται στην Ευρωζώνη, για μένα σημαντικό. Οπότε επίση και εμείς θα πούμε ναι στις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Όμως Ακόμα έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για το κείμενο. Συμφωνούμε με πολλά από τα συμπεράσματα του εισηγητή, αλλά αποκλίνουμε όσον αφορά τις λύσεις που προτείνονται από το κείμενο. Βέβαια, παρά την οικονομική ανάκαμψη, η πραγματικότητα που βιώνει ο Κοσμάκης κάθε μέρα είναι ότι συνεχίζεται η κρίση. Όλα αυτά που χάθηκαν κατά την κρίση δεν έχουν ανακτηθεί και έχει ε, επιδεινωθεί η κατάσταση εργατικής τάξης και αυτό έχει γίνει καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι αυτό το επιφανειακό, είναι ενδημικό. Πού να διορθωθεί. Δεν γίνεται με τις μικρομεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης τίποτα. Πρόκειται για το αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής αρχιτεκτονικής που έκανε το αντίθετο του σκοπομένου. Αντί να έχουμε σύγκληση, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αποκλίσεις που ριζώνουν, που αυξάνονται. Άρα έχουμε τώρα στον κατασκευαστικό τομέα ε, περισσότερες ανισότητες ε, προτείνονται τώρα ε, κάποιοι καινούργιοι θεσμοί, το εξάμεινο, το νομισματικό ταμείο που είπαμε πριν. Εμείς όμως νομίζουμε ότι για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτές τις ανισότητες χρειάζεται κάποιο πλάνο βιομηχανικό, επενδυτικό, ούτω ώστε να έχουμε κάποιον μετασχηματισμό, κάποια αλλαγή στο παραγικό μοντέλο, να έχουμε ποιοτική επασχόληση σε όλες τις χώρες μέλη και θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτούς που χτυπήθηκαν περισσότερο από την ανεργία και έτσι η ευρωπαϊκή οικονομία να πάει επομένως στην μεγάλη αλλαγή που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ένα τέτοιο πλάνο δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Και εδώ και διαφωνούμε. Γιατί το σύμφωνο σταθερότητας δεν δίνει το περιθώριο. Ούτε το πλάνο Γιούγκερ δίνει τα απαραίτητα περιθώρια. Ε, έχουμε, έχουμε συμφωνία από τις ελίτ της Ευρώπης. Αυτοί πάνε πάσο για, την, ε, για τις ανισότητες. Πιο πολύ φτωχοί, πιο πολύ πλούσιοι Επομένω, αυτοί γιατί να θέλουν να αλλάξει η κατάσταση. Επομένω, μπράβο στον εισηγητή για τι προσπάθειε του. Θα πούμε ναι σε κάποιους ε, σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, αλλά όχι στην έκθεση. Σε ευχαριστώ που τήρησε το όριο Μιγγέλ και τώρα ο Μπά για τους πράσινου. Ευχαριστίε και από εμά προ τον ε, κύριο Μπαγιέ. Όπω κάθε χρόνο είναι πια παραδοσιακή εξέταση αυτής της ε, έκθεσης, αυτής της ε, έποψης τέλος πάντων, της ανάπτυξης. Εντάξει, υπήρχαν δυσκολίε φέτος, όμως τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκητής όσον αφορά το ότι συνεκέρασε τις προτιμήσεις όλων. Ε, βέβαια, αυτό έχει το τίμημά του. Εμείς θα περιμέναμε πιο δυναμικό κείμενο, ιδίως όσον αφορά την φοροδιαφυγή, όσον αφορά την ε, τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Καλά τα είπε ο συνάδελφος από την ΚΟΕ. Θα, μπορούσαν, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αυστηροί εκεί πέρα. Το μήνυμα ποιο είναι από το κείμενο Μπαγέ ότι υπάρχει περιθώριο και χρειάζεται ε, να βρούμε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις και περισσότερη ανάπτυξη και θα πρέπει να έρθουν οι ανισότητες στην κοινωνία μας. Χρειάζονται επενδύσεις πρέπει να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε στην συνάντηση για το κλίμα στο Παρίσι. Όλα αυτά τα αποτυπώνει η έκθεση. Μπορεί εμεί να μην συμφωνούμε με όλε τι βασικέ τροπολογίε, αλλά τελικά το μήνυμα που στέλνει το κείμενο είναι αυτά τα οποία έχουμε πρεσβεύσει για το εξάμεινο. Άρα, μπράβο στον εισηγητή αποτυπώνει αυτό το οποίο έβλεπε και εμείς θα πούμε ναι στην έκθεση. Επικρίνουμε κάποια σημεία, αλλά τελικά θεωρούμε ότι μας καλύπτει το πνεύμα του κειμένου. Ε, εμείς ευχαριστούμε. Πολύ, πολύ ωραίο το ότι σήμερα έχουμε τόσο ευρεία συνένεση. Μπράβο, μπράβο, πάτε στον εισηγητή. Από το EFTD δεν βλέπω κανένα ούτε για κάποιον από το η ΕΝΕΦΑΡΑ να δευτερολογήσει ο κύριος Μπαγιέ εάν θέλει όχι όχι πρόεδρε ευχαριστώ όλους τους ε, σκιώδες εισηγητές για τη συνεργασία τους και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία πολύ ωραία θα ψηφίσουμε το απόγευμα δεν θα έχουμε καζιά, κανεί δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Επομένω, είπαμε, έχουμε 354 τροπολογίε και είπαμε ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση όσον αφορά όλου όσου έλαβαν το λόγο. Πολύ ωραία. Και τώρα. Η σκητάλη πίσω ή στον πρόεδρό μας τον κύριο Γκουαλτιέρη για το επόμενο θέμα. Και σας ευχαριστώ και πάλι. So, we move... Προχωρούμε. Πρώτη από τις δύο νομοθετικές προτάσεις. Πολύ πολύ σημαντική. Ο τίτλος είναι που θα πρέπει να το διαβάσω. Πω, πω. Θα μας φάει όλη την ώρα που έχουμε. Όχι, να μην το διαβάσω και δίνω στον εισηγητή μας τον λόγο, στον Βέρνερ Λάγκεν, για να μα προσφέρει την έκθεση του. Άρα ξεκινούμε την εξέταση έκθεση του. Βέρνερ, έχει τον λόγο. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Έχουμε ψηφίσει στις 4 Ιουλίου 2012 τον κανονισμό περί παραγόγων, η εφαρμογή ισοδυναμίας έγινε 2017 μέσω της αναγνώρισης των ΗΠΑ, 4 Μαΐου του 2017 μετά από 5 χρόνια είχαμε την πρώτη αναθεώρηση και η Κομισιόν κατέληξε στα συμπεράσματά της ε, τα οποία είναι σωστά και τα οποία δεχόμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό, κάτι το οποίο βεβαίως διευκολύνει την παρουσίαση της έκθεσής μας. Ε, θα αναφέρω τα βασικότερα ζητήματα, βελτιώνονται οι υποχρεώσεις αναφοράς, έχουμε μία μόνο δήλωση, μείωση δηλαδή της καρφιοκρατίας, το backloading καταργείται όπως είχαμε ζητήσει, μετά μιλάμε για καλύτερη ποιότητα δεδομένων και προσβασιμότητα, τα διδάγματα από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκαθάρισης επίσης ε, όσον αφορά και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλωμένους και η δυνατότητα να αναβάλουν οι αρχές την υποχρέωση εκαθάρισης βελτιώνεται. Μετά έχουμε υποχρέωση για περισσότερη διαφάνεια των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, αλλαγή της κατάταξης ε, συγκεκριμένων κατηγοριών και αυτό αφορά και τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία και επειδή είναι σωστή η κατεύθυνση δεν έχουμε κάποια ουσιαστική κριτική στην πρόταση της Κομισιόν Θέλουμε μόνο περαιτέρω διευκρινήσεις. Η έκθεση λοιπόν δημοσιεύθηκε από τη Γραμματεία 26 πρώτου και τα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν είναι αφενός το, μια βελτίωση όσον αφορά την ε, διαφάνεια, όσον αφορά τους αντισυμβαλόμενους. Μετά έχουμε την μονομερή δήλωση και βεβαίως αυτός ο οποίος κάνει την δήλωση έχει και την αστική ευθύνη. Ε, μετά έχουμε εσωτερικές συναλλαγές ομίλων που ε, δεν συμμετέχει τουλάχιστον κάποιος αντισυμβαλόμενος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πραγματική οικονομία. Μετά έχουμε παράγωγα που αλλάζουν χέρια σε χρηματιστήρια, μετά για τα συνταξιοδοτικά συστήματα θέλουμε περισσότερα κίνητρα τα οποία θα οδηγήσουν ε, σε μια αλλαγή τη κατάσταση γιατί μετά από 6 χρόνια δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδο και νομίζω ότι εδώ πέρα συμφωνούν οι συνάδελφοι. Γι' αυτό προτείναμε κάποια επιλογή που θα αυξήσει την πίεση προς την Κομισιόν και τους συμμετέχοντες. και βεβαίως ε, έχουμε και διευκρινήσεις όσον αφορά την υποχρέωση εκαθάρισης, αλλαγή της κατάταξης επιχειρήσεων, το ανέφερα, ο κανονισμός τυλοποίησης, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μετά αποτελεσματική πρόσβαση στην ε, καθάριση, το clearing και βεβαίως έχουμε ακριβώς και τα swap συναλλάγματος σε φυσική μορφή. Εδώ πέρα νομίζω ότι χρειάζεται μια παγκόσμια ρύθμιση και τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι το Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ήδη πρότεινε μια πολιτική συμφωνία η οποία δημιουργεί σε κάποια σημεία ασάφεια και περισσότερη γραφειοκρατία. αυτό θα το δούμε όταν πάμε στον τριμερή διάλογο. Κατόπιν ε, έχουμε μια σειρά συμμετεχόντων στην αγορά που πρότειναν κάποιες αλλαγές, οποίες οπωσδήποτε θα εξετάσουμε, είναι προσβάσιμες στους συναδέλφους. Όσον αφορά την δήλωση των συμβάσεων παραγόγων over the counter, τώρα δεν θέλω να τα αναφέρω όλα αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν, ε, τους ε, συναδέλφους και να υπάρξει μια σωστή εξέλιξη. Το χρονοδιάγραμμα είναι γνωστό. Μέχρι τις 28 πρέπει να παρουσιαστούν οι τροπολογίες και μετά θα πάμε σε μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε κάποια κοινά σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος ο κύριος Φονφάιστιακερ για το S&D. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Λάγκε για μια εξαιρετική έκθεση επί τη βάση μιας πολύ καλής πρότασης της ε, Επιτροπής και επί μιας σειράς πολύ τεχνικών ζητημάτων. Και οι προσθήκες του κυρίου Λάγκεν πρέπει είναι μάλλον ευπρόσδεκτες, θα αναφέρω μόνο τρεις το να συγχρονίσουμε την αναστολή της ε, υποχρέωσης εκαθάρισης είναι αυτό που έχουμε τώρα στην έκθεση του ψηφίσματος το να ασκήσουμε μεγαλύτερη θεσμική πίεση για να επιληθεί το πρόβλημα των συντάξεων θεσμοποιώντας δηλαδή τις διευθετήσεις που χρειάζονται προκειμένου να προωθήσουμε το θεματολόγιο αυτό και να προσθέσουμε και στην αρχή φραν την, ε, τον όρο διαφάνεια. Και θα μπορούσα να συνεχίσω και να αναφέρω και άλλες. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή βάση πιστεύω προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω δύο δικές μας προτεραιότητες που πρέπει πιστεύω να δούμε στενά, προσεκτικά. Ο γενικός κανόνας είναι το αντικείμενο της υποχρέωσης εκαθάρισης και να εξασφαλίζουμε στο Refit Emir να μην καταλήγουμε σε περίπτωση κατά την οποία η διασφάλιση των, της υποχρέωσης εκαθάρισης να διευρύνεται ώστε να καθυστερεί η όλη διαδικασία αδικαιολόγητα. Και δεν είμαι σίγουρος ότι μετά από τόσο χρόνο που έχουμε δώσει στην διαδικασία θα ήταν καλό να εξετάσουμε άλλη μία διετή επέκταση καθυστέρησης στην πραγματικότητα. Επομένως πρέπει να παραμείνει ευρεία η υποχρέωση αυτή. Υπάρχει και το θέμα του υπολογισμού συγκεκριμένων ορίων, κατοφλίων, όταν ε, όταν ξεκινάει να μετράει η υποχρέωση. Και η τριετία δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μαθηματικά τόσο ακριβής και ότι μειώνει και τόσο τη γραφειοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, να αναφερθώ και στο θέμα των SSPE. Ε, θέμα το οποίο πιστεύω πρέπει να εξετάσουμε από τη στιγμή που έχουμε ορίσει κάποια SSP ώστε να είναι ασφαλή και συνετά. Πρέπει λοιπόν να δούμε εννοώ πιο προσεκτικά ποια θα εξαιρούνται πιο μακροπρόθεσμα. Μια άλλη τεχνική περιοχή είναι το θέμα της υποβολής ε, ποιοτικών δεδομένων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ποιότητα δεδομένων και θα χαιρέτιζα την πρόταση της Επιτροπής να έχουμε μια έκθεση έσμα και όχι να διαγραφεί όπως προτείνει το σχέδιο του κυρίου Λάγκεν. Θα μπορούσαμε επίσης ε, στο τεχνικό μέτωπο ώστε οι identifiers των νομικών οντοτήτων να γίνουν ο κανόνας. Και με αυτά έχω ολοκληρώσει πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Keith Winmore για το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης που είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Ως μέλος της ομάδας διαπραγματεύσης επί του ΕΜΙΡ είμαι πραγματικά υπερήφανη για τα αποτελέσματα που πετύχαμε στον πρώτο γύρο και το γεγονό ότι έχει γίνει πρότυπο παγκόσμια πλέον το ΕΜΙΡ. Θα πρέπει να έχουμε τεχνικές ε, αποφάσεις που διατηρούν την προστιθέμενη αξία και ο κύριος ε, Λάγκεν με χαρά βλέπω και ικανοποίηση ότι το έχει διατηρήσει αυτό. Για τα SSP ότι πρέπει να μην κατηγοριοποιούνται ως χρηματοπιστωτικά ε, και σε σχέση με τη δουλειά που έχουμε ήδη κάνει πιστεύω ότι είναι μια θετική εξέλιξη όπως και τα swaps effects είναι επίσης προς την ίδια κατεύθυνση συνέπειας. Τώρα για την αφαίρεση της υποχρεωτικής ανάθεσης εφόσον για λόγους εσωτερικής διακυβέρνησης είναι επιθυμητό να εξακολουθήσει να γίνεται αυτό, δεν βλέπω λόγο να μην το επιτρέψουμε. Υπάρχουν και οριζόντια θέματα που μας δυσκολεύουν σε μια σειρά από φακέλους. Τα fitness check και οι εκθέσει εποπτείας αυτή τη στιγμή που υποβάλλονται. Αν δούμε ναι, συνολικά τι εκθέσεις υπάρχει ε, η αποτελεσματικότητα και η προσθέμενη αξία που επιφέρουν και το κόστος φυσικά συμμόρφωσης για τους ε, ενδιαφερομένους. Και το άκθρο τη υποβολή των εκθέσεων δεν έχει μειωθεί γιατί παρά τις καλύτερες ε, προθέσεις που έχουμε δεν έχουμε τα καλύτερα δεδομένα στο καλύτερο μορφότυπο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο οριζόντιο πλαίσιο για τη συνέχιση των εργασιών μας και ίσως θα χρειαζόμασταν μια ευελιξία σε μια τέτοια έκθεση για να ενσωματωθούν τέτοια στοιχεία για το μέλλον. Τώρα για το refit που έχουμε ξεπεράσει κάποια, από τα προβλήματα και μένοντας στο μεφύρ θα ήθελα να σημειώσω κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδυάζονται καλύτερα τα δύο κείμενα. Δηλαδή η αναστολή της ε, υποχρέωσης εμπορίας και της υποχρέωσης εκαθάρισης είναι δύο στοιχεία που θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε με κάποιο τρόπο. Και, με, οι υπηρεσίες μετά την εμπορία, ε, όπως και οι συμπίες του χαρτοφυλακίου, είναι δύο τέτοια σημεία. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε προσεκτικά τα συνταξιωτικά ταμεία και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο εισηγητής μικρής κλίμακας ε, ε, διαχειριστές χαρτοφυλακίου ώστε οι ευρωπαϊκές εντότητες να έχουν ένα ισότιμο παιχνίδι, ισότιμους κανόνες. Ω προ τον κίνδυνο που επιφέρουν τα συνταξιωτικά ταμεία και τα χρηματοπιστωτικά ταμεία ή την έλλειψη του κινδύνου που επιφέρουν στο πιστωτικό σύστημα, πρέπει να δούμε πόσο αντίστοιχε ή ομοιόμορφες είναι αυτές οι κατηγορίες. Και θα μπορούσαν να υποφελούνται από τις αντίστοιχες εξαιρέσεις με τους αντισυμβαλόμενους των χρηματοπιστωτικών είναι τα μεγαλύτερα συνταξιωτικά ταμεία που υποβάλλονται, που μάλλον που θα λάβουν ειδική μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν στην, ε, υποχρέωση εξαίρεση. Ε, καθάριση με συγχωρείτε. Και να βρούμε κάποια άλλα ελάχιστα όρια που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όμω ε, περιμένουμε ενδιαφέρον τη συνέχιση τη δουλειά μα με τον κύριο Λάγκεν. Thank For the ALDE group. ALDE. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εισηγητά για το σχέδιο του κειμένου. Η Άλτε είναι ικανοποιημένη το δρόμο που πήρε η πρόταση της Επιτροπής. Έτσι θα μειώσουμε τις δαπάνες, τις επιβαρύνσεις των παραγόντων της αγοράς θεωρούμε θετικό το σχέδιο του κειμένου έχει βγάλει από τον ορισμό τα ειδικά οχήματα εξασφάλισης. Για την τιτλοποίηση. Θα πρέπει για την αγορά της τιτλοποίησης να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία. Επίσης, είπαμε ότι οι συναλλαγές intra-group δεν θα υπόκεινται, θα ξερούνται τέλος πάντων από την υποχρέωση κοινοποίησης. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Είναι σαφές ότι τις επόμενους μήνες Ήδη τα χρόνια. Δεν θέλετε το θέμα όσον αφορά την εξαίρεση των συνταξιδοτικών ταμείων από την υποχρέωση για εκαθάριση. Ε, αυτό ότι ισχύει τώρα θα πρέπει να συνεχιστεί το πιο λογικό και έτσι οι πράγματα της αγοράς και οι εμπλεκόμενοι να μπορέσουν τελικά να βρουν μια μακρόπνοη λύση. Συγκεκριμένα τώρα. Ερωτώ τον εισηγητή αλλά και την Κομισιόν. Τι θα γίνει για αυτό το οποίο περιγραφεί με το August. Όταν έχουμε το Refit για το Mifid και όταν υπάρχει νέο νομικό καθεστώς πώς θα αποφύγουμε την αβεβαιότητα που αυτό θα δημιουργήσει στην αγορά. Χρειάζεται κάποια ταχεία λύση. Το Φραντς συμφωνούμε και επίσης θα πρέπει οι εταιρείε που κάνουν την εκαθάριση να λειτουργούν σε βάση που να αποτελεσματικότητα. Τέλος. Όσον αφορά την υποχρεωτική ανταλλαγή των περιθωρίων διακύμανσης προτείνει ο εισηγητής αυτό να περιστεί στα swaps. Θα πρέπει να φυγαμιστούμε με το τι ισχύει σε άλλες χώρες και έτσι θα πρέπει να υπάρξει θυμητός ανταγωνισμός. Άρα είπαμε ότι έτσι είναι σωστό το ότι θα μειωθούν οι επιβαρύνσεις για την αγορά. Να είναι θετική η κατάληξη και να μην υπονομεύσουμε τις αρχές που διαπνέουν τον Εμμύρ, κάτι το οποίο ισχύει παγκόσμιο. Υπάρχει κάποιος από την ΚΟΕ. Σκιώδης της ΚΟΕ. Όχι. Ο κύριος Λάμπερτς για τους πρασίνους. Καλημέρα σας. Εδώ και μια δεκαετία η χρηματοοικονομική κρίση σοβεί και θυμάμαι τι λέγαμε για τα παράγωγο που τα λέγαμε όπλα μαζικής χρηματοοικονομικής καταστροφής. Είναι θετικό ότι πολλά από αυτά τα όπλα τώρα δεν είναι αντικείμενο συναλλαγών της CCP. Αλλά γενικώ μάλλον πολλαπλασιάζονται. Μιλούμε για αγορά τεράστια. Τι είπατε κύριε Γέρτζικ ότι αυτό είναι χρήσιμο για την ανταγωνιστικότητα. Δεν είμαι και τόσο γερός. όταν άρχισα την καριέρα μου, τότε αν θυμάμαι καλά, οι εταιρείε τα πήγαν πάρα πολύ καλά και τα παραγωγά ήταν όχι υποσημείωση στην αγορά, αλλά ήταν περισμένο φαινόμενο. Και τα πήγαινε μια χαρά η οικονομία. Και πολύ θέλω να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι αυτού του είδους σώρευση όπλων μαζικής καταστροφής είναι η μόνη λύση για να προχωράει εύρυθμα η οικονομία. Και γι' αυτό το, το τι είναι, είναι απόπειρα απορρίθμισης. Κάτι εσείς μας είπατε για επιβαρύνσεις, κύριε Γερζίκ. Το λέτε εσείς επιβάρυνση, εγώ το ονομάζω προστασία. Θα πρέπει να προστατευτεί η κοινωνία από αυτά τα όπλα οικονομικής καταστροφής. Και αν μη τι άλλο θα βλέπουμε τις βασικές τάσεις, όχι, δεν θα πρέπει να κάνουμε απορρίθμιση. Θα πρέπει να νοικοκέψουμε περισσότερο την ισχύουσα νομοθεσία και το ρηφί ήταν πιο αποτελεσματικό. Δεν νομίζω ότι ωφελούν την κοινωνία αυτά τα εργαλεία, αυτά τα μέσα. Δεν λέω ότι δεν δίνουν ευκαιρίες αλλά υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτού και του να ωφελούν την κοινωνία αυτά τα μέσα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε κάποια σημεία τη έκθεση Λάγκεν. Σε μερικά άλλα σημεία έχουμε επιφυλάξει, θα θέλαμε να μα τα εξηγήσει καλύτερα. Τροπολογίε 9 και 10 που ορίζονται οι υποχρεώσεις των παρεχόντων υπηρεσίες εκαθάρισης. Θα πρέπει αυτά όλα να ξεκαθαριστούν για να μην έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων. Τώρα κάτι που πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει αυτού του είδους τα special purpose vehicles θα πρέπει να ρυθμίζονται έτσι. Μα το εξηγήσετε. 11 με 15 τροπολογίες για απλουστεύσεις σε σχέση με αντισυμβαλωμένους και τις σχετικές ε, εξαιρέσεις. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να δούμε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι εξαιρούνται και να δούμε επίσης πόσες συναλλαγές εξαιρούνται εδώ και όχι στη ΣΥΠΑ. Εδώ να διώνται ερωτηματικά. Αν είναι σωστά τα κριτήρια. Θα πρέπει να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες εξαιρέσεις. Για την αναστολή της υποχρέωσης για το clearing συμφωνούμε με τον εισηγητή. Διακόπτη ο πρόεδρος. Ω, σχεδόν σχεδόν τέλειωσε ο πρόεδρος. Ε, δεν είμαι και ο μόνος που, που, που μακρηγορώ για να μπω στις λεπτομέρειες. να υπάρχει αναστολή αυτής της υποχρέωσης όταν ξεκαθαρά δεν υπάρχει ε, κάποια εκτελεστική σύνοδο CCP μόνο εξ αυτού του λόγου να μην λειτουργεί η υποχρέωση τώρα σαν αυτά τα στελιστικά ταμεία συμφωνώ με τον Γιάκο χρειάζεται χρόνο για συμμόρφωση Οπότε θα πρέπει να είμαστε αυστηροί, να εξασφαλίσουμε ότι θα συμμορφωθούν όλοι. Και περιμένω την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα κάνουμε με τον Βέρνερ και τους άλλους οικοδησίγητες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριος να το EFTD, όχι. Ότι άλλοι συνάδελφοι, λοιπόν, τον λόγο έχει ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Μια πτυχή θέλω να αναφέρω που αναφέρθηκε ήδη για τις υποχρεώσεις ε, καθάρισης ε, και εμπορίας ε, τα οποία αναφέρονται στο μύφυρο όταν είχαμε κάνει το μύφυρο είχε ήδη εγκριθεί το ΕΜΙΡ και ως τώρα αλλάζει ο ΕΜΙΡ και πρέπει να σκεφτούμε το τι ε, θα γίνει και στην πλευρά του Μίφυρ γιατί είναι νομίζω υπαρξιακό το ζήτημα να είναι συγχρονισμένα αυτά τα δύο ε, είχαμε νομίζω και στο Μίφιτ ε, παρόμοιες συζητήσεις θα υποβάλλω νομίζω μια τροπολογία για να κάνουμε μια γέφυρα για να παρακυρίσουμε την Κομισιό να κάνει κάτι και στην πλευρά του Μηφύρ. Οπότε θα μου επιτρέψετε να υποβάλω κάποια τροπολογία τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση για να είναι συγχρονισμένα αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε λοιπόν και την Επιτροπή εδώ πέρα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Πάτρικ Πίρσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είναι σύντομος. Καλωσορίζουμε την έκθεση του εισηγητή. Είναι λογική, ρεαλιστική, εφικτή και αντικατοπτρίζει την εμπειρία του Δ. Λάγκεν στο θέμα. Είναι μια βάση για πρόοδο στο θέμα. Χαιρόμαστε για το ότι ο εισηγητής ε, δέχεται την ανάγκη αναδιατύπωση, απλοποίηση και μείωση του κόστου. Επίση θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε γρήγορα αποτελέσματα στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τροπολογίες μέσα Αυγούστου για τον ΕΜΗΡ και ειδικά το θέμα των συνταξιδοτικών ταμείων όπω ανέφερε και ένα προηγούμενο ομιλητή. Πέντε συγκεκριμένα πράγματα. Συνταξιδοτικά ταμεία. Ο τελικό στόχο είναι τα ταμεία να εκαθαρίζουν τις συμβάσεις τους ε, και να παρέχουν εγγυήσεις όπως έχουμε αποδείξει δεν υπάρχει μια μαγική λύση έχουμε ξοδέψει χρόνο ε, ένα έτος και πάνω μιλώντας ε, με τους ενδιαφερόμενους είχαμε μια ενδιάμεση έκθεση θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα λύσης θέληση υπάρχει από όλους αλλά χρειάζεται χρόνος δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε μια ημέρα. με γραμματεία της ΕΚΟΝ συμμετέχει και γι' αυτό θεωρούμε ότι η πρόταση η δική μας για τρία συν δύο χρόνια είναι απολύτως αναγκαία. Το δεύτερο είναι ο υπολογισμός ε, της εκαθάρισης για τους ε, χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλόμενους. Εμείς ε, ξέρουμε τις μικρότερες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, αλλά όλες πρέπει ετησίως να υπολογίζουν και να επιτυχνύουν ότι δεν φτάνουν στο κατόφλι που τις έξερει. Τώρα ο εισηγητής έκανε κάποιες καινοτόμε προτάσεις για να γίνει ο υπολογισμός αυτός εθελοντικός. Ε, λογικό είναι να μειωθεί αυτό αυτός ο υπολογισμός του κατοφλίου γιατί οι μεγάλε εταιρείε ξέρουν ότι θα είναι πάνω από το κατοφλί. Το θέμα είναι πώ θα ξεκαθαρίσουμε την διατύπωση για να είναι λογικό για τους μικρότερους αντισυμβαλόμενους. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει νομίζω καλύτερα. Τώρα, αναφέρθηκαν επίσης και οι προηγούμενοι ομιλητές ε, στο ζήτημα της ε, εκαθάρισης ε, και υπολογίζεται ότι και οι μικρότερες εταιρείε δεν θα πρέπει να υπάγονται σε αυτό το καθώς και οι μικρότερες εταιρείες. Αν όμως εξαιρέσουμε τις εταιρείε αυτές από τις υποχρεώσεις εγγύησης, ίσως κάνουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει κίνδυνο σε αυτές τις εταιρείε, είναι αναμφίβολο και δεν χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη του κινδύνου. Αν λοιπόν δεν έχουν αυτές τις υποχρεώσεις για παροχή εγγυήσεων, μήπως αυξάνουμε τα προβλήματα, γιατί όλοι αυτοί οι αντισυμβαλόμενοι ήδη ανταλλάσσουν τα περιθωριά τους. Έχουν σχετικές συμβάσεις ε, και θα πρέπει ακριβώς να διαπραγματευτούν τις ε, συμβάσεις αυτές και δεν βλέπουμε το πλέον έκτημα εδώ. Για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείε που δεν είναι τράπεζες, δεν είναι επενδυτικέ εταιρείε, υπάρχει ο λόγος να εξαιρεθούν για τα παραγωγά τους εάν φτάνουν στο κατόφλι. Το ίδιο ισχύει και ναι. Δεν τους διευκολύνουμε ιδιαίτερα. Ήδη έχουν σχετικά συμβόλαια. Πρέπει να υπολογίσουν ε, τα σχετικά περιθώρια και να ξεκαθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια τους και όλες οι εταιρείες που συναλλάσσονται με μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πάντα ζητούν εγγύησει. Τέταρτον, οι μονομερείς ε, αναφορές. Είναι η Νιρβάνα, είναι η Βαλχάλα, είναι ο Παράδεισος πρέπει πάντα να το εξετάζουμε και έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ο εισηγητής πάντα δηλαδή να ξέρουμε ποιος είναι τελικά υπεύθυνο για τα δεδομένα είναι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τι θα γίνει εάν τα δεδομένα που τους έχουν δώσει είναι λαθασμένα ποιος είναι υπεύθυνο, κάποιον τρόπο θα βρούμε το πέμπτον, κάποια μικρά ζητήματα, η εξαίρεση των SSP για τίτλοποιημένα στοιχεία και το Συμβούλιο εδώ πέρα συμφωνεί να εξαιρεθεί. Η Κομισιόν βλέπει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην πράξη η πρότασή μας και ίσως καμιά φορά έχει σημασία να έχουμε δίκιο από το να είμαστε συνεπείς. Οπότε βλέπουμε που πάει η συζήτηση. AIF ε έχουν γίνει πολύ σωστές ε, προτάσεις επίσης για συμβόλαια μελλοντική εκτέλεσης ε, συναλλάγματος απολύτως σωστό και χαιρόμαστε που το ανέφερε το Κοινοβούλιο ο κ. Φέρμπερ είπε κάτι πως θα συγχρονίσουμε την ΕΜΙΡ και το ΜΙΦΙΤ είναι περίπλοκο το ζήτημα θα το μεταφέρω στους συναδέλφους που είναι αρμόδιοι για το ΜΙΦΙΤ και προτείνω να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να βρούμε μια προσέγγιση και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα νομίζω στην πράξη στις αγορές αν συμφωνεί και ο κύριος Φέρμπερ ευχαριστώ και για αυτά τα οποία είπατε και χαίρομαι ακριβώς ε, που θέλετε να συζητήσουμε το θέμα Βέρνερ ακούσατε πολλά σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις σας το θέμα μας απασχολεί από το 2009 ε, μετά από το Pittsburgh το 2009 είναι επιτάπητος και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι είναι εδώ η κυρία Σουίνμπερν τότε ήταν εξαιρετική σκιώδης εισηγήτρια και βεβαίως απαραίτητη γιατί έχει εμπειρία στον κλάδο οι προτάσεις ε, έγιναν, τις σημειώσαμε υπάρχουν τα βασικά θέματα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με τα κατά μία. θα το συζητήσουμε. Εξαιρέσει για τις μικρότερες εταιρείε και ένα πιθανό κατόφλι, θα το δούμε όπως είπε και ο κύριος Πίρσον. Το άλλο είναι ακριβώ ε, το πώς θα καθορίσουμε την υποχρέωση αναφορών ε, και το άλλο είναι όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν από την προθεσμία μέχρι την ε, Μίφιντ και εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν δούμε τις τροπολογίες να προχωρήσουμε γρήγορα χωρίς πάρα πολλές ε, συναντήσεις ε, σκιωδών όπως γίνονται τώρα στον τομέα της ενέργειας εντός της προθεσμίας και να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τον επικοδομητικό διάλογο που κάνουμε με τον κύριο Πίρσον από το 2010. Ευχαριστώ. Thank you, Bernard. Are you already... Ευχαριστούμε, Βέρνερ. Η προθεσμία λοιπόν για τις προθεσμίες είναι 28 Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα, 19 Μαρτίου εξέταση τροπολογιών, 8 Απριλίου ψήφος. Νομίζω ότι είναι ένα συνολικά σωστό χρονοδιάγραμμα. Και προχωρώ στο επόμενο σημείο, πάντα εμμύρ. Διαδικασίες που σχετίζονται με την έντριση των, έγκριση των κεντρικών αντισημαλωμένων. Η κυρία Χύμπνεα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με αυτήν την δήλωση που ακούμε συχνά στις εκθέσεις μας ότι δηλαδή όλα αυτά έγιναν επί τη βάση μιας πολύ καλής προτάσεως κομισιών. Προτείνεται λοιπόν τροποποίηση της εποπτείας με πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. και των ε, συμβαλωμένων των τρίτων χωρών που εκπροσωπούν δηλαδή αγορές που είναι σημαντικές για τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια αναλογικότητα και εγώ θα έλεγα ότι είμαι υπέρ της γενικής κατεύθυνσης την οποία δείχνουν οι προτάσεις της Κομισιόν. και θα αναφέρω κάποια ζητήματα που θεωρώ πολύ σημαντικά σε αυτήν την πρόταση. Σε πολλά από αυτά συμφωνώ με την Επιτροπή, σε άλλα αποκλίνω κάπως. Καταρχάς τη διαδικασία μη αναγνώρισης κάποιου τρίτου CCP που είναι ένα είδος εγγύησης αν θέλετε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά αλλά χρειάζονται πιο σαφή κριτήρια. Με ποιο τρόπο αρνούμαστε την αναγνώριση CCP της χώρας. Ε, κατά την άποψή μου το σύστημα που προτείνεται αυτή τη στιγμή ε, είναι κάπως ε, διακριτικής προσέγγισης, θα έλεγα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει η όποια ε, απόφαση λαμβάνουμε να βασίζεται στις ενδείξεις, στις αποδείξεις, να είναι πιο αντικειμενική. Το σύστημα πρέπει να είναι αξιόπιστο και επομένως πρέπει να βασίζεται επί των αποδεκτικών στοιχείων και πρέπει να εξασφαλίζουμε στο μέτρο του δυνατού ότι οποιαδήποτε απόφαση κατάσταση δεν έχει περισσότερο αρνητικό παρά θετικό αντίκτυπο επί των Ευρωπαίων εταίρων. η ανάλυση ΕΚΤ ΕΣΜΑ σχετικά με τις υπηρεσίες καθάρισης ε, και την άρνηση αναγνώρισης αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ε, συνδιαλλαγής. Δηλαδή αν έχουμε ρέπος, αν έχουμε νομισματική μεταφορά ή άλλου είδους συνδιαλλαγές Ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να εισαγάγει κάποια στοιχεία ώστε να αντισταθμίζεται αυτή η άρνηση αναγνώρισης, μια δηλαδή μεταβατική περίοδος για πελάτες και για μέλη. Και ίσως η Κομισιόν επίσης ε, με την εκτελεστική πράξη θα μπορούσε να επιμείνει λίγο περισσότερο στις υφιστάμενες ε, συμβάσεις. Γιατί μάλλον αυτό το στοιχείο είναι από τα πιο προβληματικά σε, στην περίπτωση δηλαδή μη, ε, άρνησης αναγνώρισης CCP. Επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα άρνησης μόνο για την υπηρεσία εκαθάρισης και όχι για το σύνολο του αντισμαλωμένου. Και εδώ θα μπορούσε να εισαχθεί μια κάποια αναλογικότητα το οποίο θα καθιστούσε αυτό το στοιχείο πιο ευθυγραμμισμένο με τη διαδικασία που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, με την παροχή ή μη παροχή έγκρισης. Επίσης υπάρχει το θέμα της οργάνωσης της ΕΣΜΑ για την εποπτεία. Χρειαζόμαστε μια δομή που να μην είναι απολύτως ανεξάρτητη από το υπόλοιπο της ΕΣΜΑ και να συνδέεται δηλαδή με τον υπόλοιπο φορέα που να επιτρέπει και μια κάποια οριζόντια συζήτηση εντός της ΕΣΜΑ Ίσως λοιπόν μια ιστορική επιτροπή της ΕΣΜΑ θα μπορούσε να έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας ε, των αντισμαλωμένων και των ευρωπαϊκών και των τρίτων χωρών και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να παραμείνει αναξαρτήτως της ε, επανεξέτασης γιατί αυτά απορρέουν από το άρθρο 41 του κανονισμού της ΕΣΜΑ και εδώ προτείνω λοιπόν ότι η αρμοδιότητα θα έπρεπε να είναι και επί των ευρωπαϊκών και επί των CCP ε, των τρίτων χωρών. Και η τρίτη πτυχή είναι η κεντρική τράπεζα έκδοσης και ο ρόλος της εδώ. Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να ενέχονται σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων έχει αντίκτυπο επί της νομισματικής πολιτικής. Το πεδίο της αρμοδιότητας λοιπόν των κεντρικών τραπεζών φαίνεται να είναι καλά ορισμένο στην πρόταση, αλλά και εδώ ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια σαφέστερη περιγραφή του ορίου της αρμοδιότητας και σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο θα πρέπει να παρεμβαίνει. Να παρεμβαίνουν. Και πρέπει να καλύψουμε και τις περιπτώσεις και τις οποίες θα είχαμε αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ ΕΚΤ και ΕΣΜΑ. Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε διάφορες ιδιαιτερότητες αλλά μπορεί να έχουμε και περιπτώσει κατά τι οποίε χρειαζόμαστε ταχείες αποφάσεις και μία αρχή, έναν φορέα που θα πρέπει να είναι επικεφαλής. Δεν είναι τόσο εύκολο η ΕΣΜΑ είναι ένας οργανισμός και δεν είναι ένας θεσμικός φορέας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα είχα λοιπόν την τάση να πάμε προς ένα μηχανισμό εξήγησης της συμμόρφωσης, δηλαδή ότι θα πρέπει να δικαιολογείται η οποιαδήποτε απόκληση προς τη γνωμοδότηση της ΕΚΤ. Αλλά εδώ ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και τη βοήθεια ενός συνέδελφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διατυπώσουμε την πρόταση αυτή κατά τρόπον ώστε να μην αφήνει καμία αμφιβολία. Το πρώτο τελευταίο που θέλω να πω αφορά στην μετάβαση προς το νέο καθεστώς της χώρας είχαμε αποφάσεις ε, υπό το προηγούμενο καθεστώς ισοδυναμίας όπου έχουν αναγνωριστεί δηλαδή κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι σε 15 διαφορετικές ε, ε, χώρες. Κράτη στην ουσία. Αρμοδιότητος δηλαδή των κεντρικών του τραπεζών για να δούμε σε ποια κατηγορία θα πρέπει να εμπίπτουν αυτοί οι CCP θα χρειαστεί δηλαδή ε, μια στενή αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και θα πρέπει από κοινού εδώ να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. και να αναφερθώ και σε αυτό το θέμα της ε, συνεργασίας για την εποπτεία. Δεν είναι ε, επαρκές απλώς να υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων ή στο πλαίσιο ενός κανονισμού. αλλά στο μέτρο που μπορούμε νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις συνδίκες καλής συνεργασίας μεταξύ ΕΣΜΑ και των εκπροσώπων της ε, Κεντρικής Τραπέζας αλλά και των εκπροστόπων της ε, ρυθμιστικής αρχής της τρίτης χώρας. Χρειάζονται λοιπόν ε, μνημόνια συνεννόησης και πρωτόκολλα ακριβή και συγκεκριμένα προκειμένου να αναπτύξουμε μια καλή σχέση συνεργασίας σε καθημερινή βάση. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε, να ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο καλής συνεργασίας, διότι θα έχουμε και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης όπου θα χρειαζόμαστε, ξαναλέω, ταχεία διαδικασία λήψη απόφασης και μια τέτοια καλή συνεργασία είναι απαραίτητη σε εκείνη την περίπτωση. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα νότα. Τώρα θα μιλήσω ως ε, της ε, των σοσιαλδημοκρατών. ευχαριστώ την έκθεσή σας. Όπως επίσης ε, και το ότι ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της ε, Κομισιόν, η οποία συμφωνώ μαζί σας είναι πολύ ισορροπημένη. Είμαστε πεπισμένοι ήδη, έχουμε πει ότι μια αναθεώρηση της ε, εργασία ε, αναγνώρισης ε, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και των τρίτων χωρών απαιτείται ε, εν ώψη του Brexit αλλά και του ότι έχουμε πλέον υποχρεωτική εκαθάριση και για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά για να προχωρήσουμε γρήγορα και καλωσορίζω επίσης το ότι η έκθεσή σας ε, ε, συνετάχθη πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεί νομίζω μια καλή βάση συνεργασίας για να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους. Αναφέρατε κάποια πράγματα και θα ακολουθήσω και εγώ την ίδια σειρά λίγο πολύ. Καλωσορίζω, όπως είπα, το ότι σε γενικές γραμμές είμαστε, θα έλεγα, κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να τα συζητήσουμε και στην ομάδα μας, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια βάση συνένεσης. Συμφωνούμε για την επιλογή σας να διατηρηθεί μια συμμετρία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κεντρικών αντισυμβαλουμένων τρίτων χωρών. Αντιλαμβανόμαστε ότι οπωσδήποτε είναι κάπως επώδυνο αλλά χαίρομαι που επιβεβαιώνεται αυτή την προσέγγιση για την συγκεκριμένη πρότασή σας για την Εποπτική Επιτροπή είναι οπωσδήποτε μια επιλογή και αυτή και συνδέεται με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Αξιών και Αγορών ε, γιατί βεβαίως το Κοινοβούλιο ε, είναι το αρμόδιο όπως ήταν και στις άλλες προτάσεις οπότε θέλουμε να το δούμε αυτό για τη διαδικασία για την αναγνώριση ορίζω αυτό το οποίο είπατε την αξιολόγηση δηλαδή κόστους κόστους-οφέλους την βιωσιμότητα την δυνατότητα να διακρίνουμε μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών εκαθάρισης και την ε, μεταβατική περίοδο όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία και συμφωνούμε με την πρόθεση που εκφράζεται σε αυτές τις ε, τροπολογίες για την Κεντρική Τράπεζα Έκδοσης ε, μία επιλογή είναι και η λύση που προτείνεται. Όπως είπατε, ε, δεν είναι αυτό ακόμα στην εκθεσή σας, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε κάποιους μηχανισμούς, μια διαδικασία α, συμμόρφωσης ή εξηγήσεων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, αλλά είμαστε ανοιχτοί στον εξετάσουμε το θέμα για το καθεστώς ε, τρίτης χώρας όπως είπατε για το θέμα της ε, συγκρίσιμης ε, συμμόρφωσης και καλό είναι το ότι δεν αμφισβητούμε τις υφιστάμενες αποφάσεις ισοδυναμίας βεβαίως δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την Ένωση από το να ε, έχει ένα τέτοιο μηχανισμό. Γι' αυτό ακριβώς θα εξετάσουμε την αναγνώριση. Ίσως βεβαίως η περίοδος να μοιάζει σύντομη. Θα το εξετάσουμε, αλλά αν το υπολογίσει κανείς ε, είναι μεγαλύτερη η περίοδος από ό,τι φαίνεται, γιατί πρέπει το εγκρίνουμε να τεθεί ενισχύ, πράξη ε, κατεξουσιοδότηση. Ε, θα περάσουν κάποια χρόνια δηλαδή αλλά θα το εξετάσουμε και οπωσδήποτε θα κοιτάξουμε με ε, ε, οποιονδήποτε τρόπο για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση λαμβάνοντας πάντα υπόψη ε, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Νομίζω ακριβώς θα σκεφτούμε το πώς θα ξεκαθαρίσουμε ότι δεν σκοπεύουμε να ρυθμίσουμε εμεί συζητήματα Αμερικανών αγροτών και γεωργικών παραγόγων που για αυτή τη στιγμή. Οπότε θα το δούμε. Γνωρίζουμε βεβαίω πως οι συνδυασμοί των διαφόρων πτυχών και παρομοίες συμμόρφωσης μπορούν να επιτρέψουν στην Ένωση να ενισχύσει και να βελτιώσει τα εποπτικά της εργαλεία από την άλλη βεβαίως διατηρώντας ε, το υφιστάμενο πλαίσιο συμφωνιών που έχει μέχρι στιγμής επιτύχει. Νομίζω λοιπόν περιλαμβάνοντας βεβαίως, και το θέμα το οποίο αναφέρατε για την εποπτική συνεργασία νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια ευρεία κοινή βάση. Βεβαίως υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε συνεργασία πάντα με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Οπότε η ομάδα μας ε, θέλει να επιτύχει ακριβώ μια συνένεση και να προχωρήσουμε γρήγορα. Οπότε τώρα περνάω στην Κέι Σουίνμπορν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Τανούτα Χούμπνερ για την δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι βελτιώνει την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Η οποία είναι βέβαια μια πολύ καλή αρχική βάση δουλειάς. Θα μείνω σε τρεις περιοχές. Καταρχάς, η σαφής διαδικασία λήψης απόφαση της νέας δομής, η πρωτοκαθεδρία της Κεντρικής Τράπεζας Έκδοσης που παραμένει στο κείμενο και η ισοδυναμία των τρίτων χωρών. Και μετά θα δούμε και την πολιτική μετεγκατάσταση Για την Επιτροπή Εποπτεία και το νέο σχεδιασμό τη. η μετακίνηση που προτείνεται μου έδινε μια πρώτη εντύπωση ότι αυτό είναι σαν ε, συλλογικός φορέας κολέγιο, αν θέλετε, των CCP. Η ανησυχία μου εδώ είναι ότι ίσως να μην δίνει την μονιμότητα, τη σταθερότητα ενός σώματος, ενός φορέα με τον οποίο θα πρέπει να έχουμε οποιαδήποτε θεσμική σχέση. Και με το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, η ΕΣΜΑ δεν θα πρέπει να αποτρέπεται από αποφάσεις εποπτείας που θα έπρεπε να μπορεί να παίρνει. Θα πρέπει να είναι σαφής λοιπόν η, η ιεραρχία του ποιος είναι υπεύθυνο σε περίπτωση διαχείρισης κρίσης και σχετικών αποφάσεων. Επίσης μπορούμε να αποφεληθούμε τη αφήνεια διαδικασίας αποφάσεω για την αναγνώριση ε, CCP τρίτων χωρών. Θα είναι απλά ο πρόεδρος της Επιτροπής που θα έχει την ε, αρμοδιότητα της απόφασης ή άλλοι εποπτικοί φορείς άλλων φορέων εκαθάρισης. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιη πώς θα είναι αυτή η αλλη εποπτικη φορεις αλλων φορεων εκαθαρισης δεν ειμαι απολυτα αρχαία η αρχιεκτονική της εκπροσώπησης των ε, CCP. Με την ε, Κεντρική Τράπεζα Έκδοσης εξακολουθώ να έχω σημαντικές ανησυχίες. Όπως βλέπουμε στην ε, έκθεση της Κομισιόν, δίνουμε το βέτο δικαίωμα ανησυχηρίας στην Κεντρική Τράπεζα Έκδοσης. και στο πεδίο των προϊόντων και στα μέλα της εκαθάρισης αλλά το να δώσουμε το βέτο σε μία μόνο κεντρική τράπεζα όταν ε, εκπροσωπούμε παγκόσμιους φορείς είναι ένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη τη σημερίζεται και η Αμερικανική ε, Κεντρική Τράπεζα. Οτιδήποτε παρεμποδίζει την δυνατότητα ενός CCP να διαχειριστεί τις συνδιαλλαγές του, τον περιορισμό των περιθωρίων του ή τη διαχείριση των περιθωρίων του, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Νομίζω λοιπόν ότι η τροπολογία 67 εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αναγνωρίζεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να περιορίζει τη δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας Έκδοσης σχετικά με την κατά πόσον εμπίπτει η κάθε περίπτωση το ΕΜΗΡ ή όχι. Επίση, όταν μιλούμε για το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας Έκδοση σε συγκεκριμένες τρίτες χώρες και εδώ υπάρχουν ανησυχίες και πρέπει να αποσαφενίζουμε ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο ε, παραχώρηση ρευστότητα σε τρίτη χώρα CCP. Δηλαδή οποιοδήποτε swap line που έχει ενεργοποιηθεί από ε, CCP του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια κατάσταση Brexit θα εγγυάται πλέον από την Τράπεζα της Αγγλίας. Το οποίο θα ισχύει και για την ε, Fed, για την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή πρέπει να δούμε κατά πόσον η εγγύηση παρέχεται από άλλη τράπεζα έκδοσης ή από την ίδια την οντότητα. αλλά αυτή η οντότητα σε σχέση με την χώρα στην οποία ανήκει, έχει δικαιοδοσία. Η ισοδυναμία CCP ε, όταν την εξετάζαμε για τι Ηνωμένε ήταν ε, αναβάση χώρα και όχι οντότητα και μα πήρε και τρία χρόνια εκείνη η δικασία. Τώρα για να έχουμε αναγνώριση οντότητο στην ουσία θα έπρεπε να, ε, το εξετάζουμε ως ένα θέμα ισοδυναμίας τρίτης χώρας. Δηλαδή είναι ένα θέμα συσχετισμού ε, ε, εταιρεία, οντότητος και χώρας. Είχαμε μακροσκελή συζήτηση εχθές με την CFTC όπου μας εξήγησαν τι σημαίνει για εκείνους ο όρος deference και δεν σημαίνει διπλή εποπτεία, σημαίνει συνεργασία και σημαίνει ότι πραγματικά εμπιστεύεται κανείς την εποπτεία που θα παράσχει, που θα εξασφαλίσει ο άλλος εταίρος ή τρίτη χώρα. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υποδαβλίσουμε αυτόν τον τρόπο της οικονομικής συνεργασίας που είναι παγκόσμια. Επομένως η, συγκριτική συμμόρφωση που αναφέρουμε εδώ είναι σημαντική και θα χρειαστούμε περαιτέρω προσπάθειες να αξιολογούμε την ε, συμμόρφωση αυτή γιατί υπάρχει μια έλλειψη σαφήνεια στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Υπάρχουν κάποια κεντρικά σημεία του πώς αξιολογεί κανείς ε, CCP τρίτης χώρας. Ακούσαμε αρκετές ανησυχίες για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν αυτά στην πράξη και νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Πάντως δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περαιτέρω για την πολιτική μετεγκατάσταση, αν ακούσαμε καλά, αλλά είναι σημαντικό να δούμε τι ενδείξεις, τι σημάδια διαβιβάζουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Πάντως, εγώ χαιρετίζω την ε, ε, αναγκαιότητα της ΕΣΜΑ να προχωρήσει σε μια ανάλυση κόστος ωφέλους προτού εφαρμόσει το οτιδήποτε και η Κομισιόν θα πρέπει να βασιστεί σε εκτελεστική πράξη επί τη βάση της ε, σύστασης της γνωμοδότησης που θα δίνει η ΕΣΜΑ. Και επίσης θα μας χρειάζεται ε, ένα, μια περίοδος μεταβατική. Τα swaps, τα repos και τα λοιπά δεν πρέπει να αποκλίνουν από το προφίλ του κινδύνου τους γιατί πολλές επιχειρήσεις έχουν αντίστοιχο προϊόν στην άλλη πλευρά. Δηλαδή σε ένα swap όταν έχουμε ορίσει το, το ισοδύναμο ή αν θέλετε το συμμετέχον προϊόν που είναι ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, τι θα κάνουμε με το εξωτερικό, με τις τρίτη χώρα. Επομένως χρειάζεται μια προσεκτική προσέγγιση. Ευχαριστώ όμως την εισηγήτρια στην προσπάθεια που έχει καταβάλει μέχρι τώρα και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα το σχέδιο. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Ω, βέβαια. θα πρέπει να εξηγήσουμε την επιχειρηματολογία μας που μας οδηγεί σε επιφυλάξεις που διατύπωσες. Πέτερ Γέζεκ. Ρομπέρτο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την συγκεντρία για το σχέδιο της ε, έκθεσης και για τη συνεργασία της σε όλη τη διαδρομή. Τρόσον αφορά την ε, έκθεση η συγκεντρία έχει κατελήξει ένα ισορροπό κείμενο, έχει στηριχθεί στις προτάσεις Επιτροπής, έχει επεξεργαστεί για λεπτομέρειες. Για να σας πω τώρα μερικά σημεία και να δούμε τι μπορούμε και τους επόμενους μήνες να συζητήσουμε όσον αφορά την εποπτεία των συζητήσεων σε επίπεδο ένωσης. Είναι θετικό αυτό που κάνει η συγγήτρια να προσπαθεί να προσθέσει τα της εκτελεστικής συνόδου. Επίσης νομίζουμε το τροποποιημένο αυτό πλαίσιο προσθέτει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Πάντως, επίσης να αναγνωρίσουμε το ότι όλα αυτά έχουν σχέση και με την τροποποίηση και εξολόγηση της ΕΣΑ Θα δούμε με την διακυβέρνηση ε, για την υπόθεση των CCPs, με σύνοδο, γιατί νομίζω ότι έχουμε τώρα κάποιες άλλες ε, επιλογές να τις μελετήσουμε για να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Επίσης όσον αφορά τις διευκρινήσεις της ηγήτριας είναι σωστό να έχουμε αυτά τα κριτήρια για το σε ποια κατηγορία θα εμπίπτουν τα CCP κάθε χώρας και να δούμε πώς θα ρυθμιστεί η ισοδυναμία. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και η απόφαση να μην στηρίζεται σε πολιτικά κριτήρια, αλλά σε αντικειμενικά κριτήρια και τεχνικά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ευρώπη. Και έτσι θα πρέπει να διαμορφώσουμε την υποπτία των CCP. ακριβώ όπως είπαν διάφοροι συνάδελφοι. Έχουμε συμφωνίες με διάφορους σε όλο τον κόσμο. Και αλλαγέ που θα κάνουμε στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τα όσα έχουμε συμφωνήσει με τους εκτός Ευρώπης εταίρους μας. Επίσης, θα πρέπει να διαχειριστούμε και να νοικοκυρέψουμε την εποπτεία μας. Να δούμε τι γίνεται με την εποπτεία στον υπόλοιπο κόσμο και πώς γίνεται με τον πιο στο τρόπο η δουλειά. Ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Γουαλτιχέρη, γιατί είναι το λόγο στον κύριο Λάμπερτς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την Τανούδα για αυτή την μεστή έκθεση συμφωνούμε ότι θα πρέπει τα CCP να έχουν πιο αποτελεσματική, πιο στεγανή εποπτεία. Είναι συστημικό στοιχείο του χρονοτολογικού συστήματο. Είναι πολλά και περισσότεροι κίνδυνοι. Ε, και γι' αυτό χρειάζεται να είναι πανευρωπαϊκή η προσέγγιση. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον κανονισμό ΕΣΜΑ. Χρειάζεται εμπειρογνωμοσύνη και στο τοπικό επίπεδο και να ξέρουμε ότι οποιαδήποτε εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται όπως πρέπει. Συμφωνώ ότι το να εμπλακούν οι κεντρικές τράπεζες ε, θα πρέπει αυτό να το ρυθμίζουμε πέρας πρώτες κομισιόν για να υπάρχουν κάποια μέτρα και νομοθετικά αλλά αυτό ίσω είναι περίπλοκη διαδικασία. Καλά, να βοηθήσουμε με δικέ μας προτάσεις. Και συμφωνούμε με την Τανούτα. Με αυτό που λέει δηλαδή η Κομισιόν, ότι το σημερινό καθεστώς στηρίζεται υπερβολικά στην υποπτή των τρίτων χωρών. Αυτό όμως δεν ε, ε, ταιριάζει ε, σε κάποια CCP που είναι συστηματικής, συστημικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει στο πρώτο επίπεδο να δούμε ε, σε ποιο επίπεδο θα κατατάσσονται οι διάφορες ε, CCP Ιστορική Επιτροπή αντί για το τι προβλέπει τώρα ο κανισμός ΕΣΜΑ πέραν του τι άλλες αλλαγές θα γίνουν. Όμως δεν έχουμε πιστεί ότι αυτή η πρόταση θα διευκολύνει τις αποφάσεις. Γιατί μπορεί να προσβληθεί δυνάμει του έσμα οποιαδήποτε απόφαση. Και άρα θα πάσχει νομικά αυτή η λύση. Να δούμε τι άλλες λύσεις υπάρχουν και έτσι να μην μπλέξουμε με περισσότερη γραφειοκρατία και επίσης να είμαστε συμβατοί με οτιδήποτε μέλουσα μορφή της ΕΣΜΑ στα πλαίσια της αξιολόγησης της EAS. Μπράβο, μπράβο στην Τενότα και ελπίζουμε η θέση μας τελικά να είναι αξιόλογη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο κ. Γκολτιέρη. Δεν βλέπω άλλον σκιώδη ηγητή να το λόγο. Και άρα δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πίρσον. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόταση που ορίζει το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα μέσα, για αυτούς τους φορείς, γιατί χρειάζεται η ρύθμιση αυτή να ξεκάθαρα για να ωφεληθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Χούμπνερ για την έκθεση, για τις ε, προτινόμενες τροποποίησεις της δικής μας πρότασης είναι εύστοχες, είναι ευφύς ε, μεταβολές και άρα είναι μια πολύ καλή αφετηρία για το μέλλον. Η πρόταση της Κομισιόν ε, είναι ε, απαραίτητη ούτως ώστε να βελτιωθεί η εποπτεία των ΣΥΣΥΠΗ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι θέλουν δηλαδή να μπουν στις αγορές της Ευρώπης και να προσφέρουν εδώ τις υπηρεσίε τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι για να έχουμε καλύτερη εποπτεία. Τρεις παρατηρήσεις. Θέλω να πάρα πολύ θετικό το ότι η συγκήτρια συμφωνεί με όλα τα βασικά σημεία της πρότασής μας. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη ότι θέλει μεγαλύτερη εμπλοκή των κεντρικών μας τραπεζών στην υποπτία. Και επίσης συμφωνεί θα πρέπει να δούμε πώς όλες οι συζητοί ευρωπαϊκές και μη λειτουργούν στην Ευρώπη. Οι κεντρικές τράπεζες είναι υπεύθυνες για την νομισματική πολιτική, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ρευστότητα, πληρωμές, ε, και οι ρυθμιστικές αρχές των ε, χρηματαγορών δεν μπορούν χωρίς τις σχετικές τράπεζες να κάνουν μόνες τους την εποπτεία. Δεν υπάρχει στη, στη γη καμία χώρα που αυτό να είναι εφικτό. Θα λάβουμε όπως αυτά που είπε η κυρία Χούμνερ για να δούμε τι γίνεται με το βέτο, πώς μπορεί να δουλέψει καλύτερα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Δεύτερον, θετικό ότι θέλει να χωρίσει τις μη ευρωπαϊκές ε, σε δύο κατηγορίες, συστημικές και μη συστημικές. Αυτό έχει αναλογικότητα, ε, αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που ίσως εγκυμονούνται για το σύστημά μας και όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, θα βοηθήσει αυτός ο μηχανισμός ε, συμμόρφωσης. Και έτσι τα πράγματα θα ξεκαθαριστούν ίσως περισσότερο. Έτσι θα εξασφαλιστεί το ότι το σύστημα θα αποτελέσει βελτίωση των σήμερα ισχυόντων και θα βοηθήσει και τις άλλες χώρες. Επίσης, στην Ιταλική λέει ότι βασικό πρόβλημα των όσων σήμερα ισχύουν για τις ε, σημαντικές εισηπητήρες των χωρών που δρούν στην Ευρώπη είναι ότι το σύστημα είναι αδύναμο και στηρίζεται περισσότερο στις αρχές των τρίτων χώρων, περισσότερο πόσο θα έπρεπε. Και είναι σωστό ότι οι αγορές ε, για να είναι σταθερές στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίζουν να διέπονται από το κοινωτικό δίκαιο, από ρυθμιστικές αρχές ε, και θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Οπότε και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρυθμιστικές αρχές της ε, Ένωσης οπωσδήποτε και συμφωνούν. Πώς θα μπορούσε να μην ισχύει αυτό. Ναι, ναι, πολλά λέγονται. Κυρίως από ε, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά όπως μου λένε οι συνάδελφοι, αυτά όλα είναι κάτι σαν αυτά που έλεγε ο Σέξπιρ, ότι η Γερτρούδη γκρίνιαζε γκρίνιαζε και ξαναγκρίνιαζε και επαναλάμβανε κάτι. Αλλά τελικά είχε κολλήσει σε κάτι για το οποίο είχε δίκιο. Επομένως, ελπίζουμε ότι τελικά να μείνουμε, να είμαστε σταθεροί στη γραμμή μας, θα κατασυγάσουν οι διαμαρτυρίες αυτές. Επίσης υπάρχει και το θέμα του αν θα αφήσουμε να προσφέρουν όλες ή μόνο κάποιες υπηρεσίες τα CCP αλλά ίσως όχι αν διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικό αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα λαμβάνεται αυτή η απόφαση ποιο θα είναι το κόστος, τι θα γίνει με τις συμβάσεις περίοδοι προσαρμογής και τελικά αυτό που διακυβεύεται είναι η σταθερότητα των δικών μας αγορών και του δικού μας νομίσματος. Άρα για τίποτα απόφασή μας θα πρέπει να υποβληθεί σε εσά και στο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας χωρίς να ακούσουμε εσά και το Συμβούλιο. Για να τα ξεκάθαρα σας το λέω. Η κυρία Σουίνμπερν μίλησε για ισοδύναμες ε, αποφάσεις ή αποφάσεις τέλος πάντων ισοδυναμίας. Τι γίνεται όμω με την νομοθεσία και την εποπτεία άλλων χωρών. Όμω η πρότασή μα δεν αφορά αυτό, δεν αφορά την ισοδυναμία. Αφορά το πώ θα υποπτεύσουμε συγκεκριμένε εταιρείε από τρίτε χώρε που έρχονται στην Ευρώπη για να συναλλαγούν με τι εταιρείε μα και με του πολίτε τη Ένωση. Οπότε και εγώ σα επιβεβαιώνω ότι από όσο γνωρίζω η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει τις αποφάσεις της Καμία αλλαγή στο δίκαιο των τρίτων χωρών. Καμία αλλαγή στο ΕΜΙΡ ούτε στο κλίμα συνεργασίας με τις ε, ρυθμιστικές των χωρών. Ας γίνει ανθιόρυση αυτών των αποφάσεων αφού εγκριθεί το παραγγείμενο πρόεδρο όπως είπατε. Πρώτα, πρώτα όμως να τεθεί σε εφαρμογή. Και μετά θα έχουμε έξι μήνες για μια κατεξουδότηση πράξη. Οπότε τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει για αυτή την πράξη να τοποθετηθούν και μετά χρειάζονται 12 μήνες ώστε η εξουδότηση πράξη να τεθεί σε ισχύ και πρέπει να δούμε κατά πόσο χρειαστεί η περίοδος προσαρμογής. Ε, εγώ τότε θα έχω πάρει σύνταξη, σας, το υπόσχομαι. Σας δίνω το λόγο μου. Τέλος. Με μεγάλο ενδιαφέρον μελετούμε αυτά τα οποία είπε η εισηγήτρια για τη διακυβέρνηση για το ΕΣΜΑ. Μέα κούλπα, εγώ φταίω, γιατί εγώ κάθισα και έφτιαξα το σχέδιο κειμένου. Τι να πω, τι θα πω στη γυναίκα μου, έκανα ό,τι μπορούσα. Όμω αυτά που λέει η είναι απλούστερα, καλύτερα, αντικατοπτρίζει το τι ισχύει για την κεντρική τράπεζα, καλύπτει όλα τα σχόλια. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα ο κανονισμό ΕΣΜΑ. Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό άσχετα με την ε, αξιολόγηση ΕΣΑ. Τέλος. Μπράβο στην εισηγήτρια για τόσο από την εποπτεία των CCP. Υπάρχουν βέβαια περιπλογές με τα κρατη Και αν ε, η ΕΣΜΑ κάποιος άλλος ή περισσότερε αρμοδιότητε, αυτό σημαίνει ότι θα τι έχουμε πάρει από κάποιον άλλο αλλά το ζουμί τη πρότασή μα, αλλά και τη ηγετρίας είναι το ότι τελικά το σύνολο θα είναι πιο καλό από τα μέρη του. Άρα, περιμένουμε να μας ε, στηρίξει το Κοινοβούλιο και έτσι να μπορέσουμε με επιτυχία να αντικινηθούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πίρσον. Ντανούτα. Σύντομα κύριε Πρόεδρε γιατί τρώμε τον χρόνο της επόμενης έκθεσης. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους ε, την Κομισιόν. Ε, θα έχουμε πολλές συζητήσεις. Έχουμε αρκετό χρόνο πριν την προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα έχουμε και τις συναντήσεις των σχεδόν. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Πρέπει βεβαίως ε, η διαδικασία λήψη αποφάσεων να είναι ομαλή. Γιατί αυτή είναι νομίζω συνήθως η αδυναμία των ευρωπαϊκών προτάσεων στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Και πρέπει ακριβώς ε, να δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση όσον αφορά την νομική ασφάλεια. Γιατί όπως αναφέρθηκε αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα, αξιόπιστο και με νομική βεβαιότητα. Ελπίζω λοιπόν να διατηρηθεί αυτό το πνεύμα σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει σαφής ε, πολιτική στήριξη για ένα κείμενο το οποίο όπως είπε και η Κομισιόν έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης της ε, Κομισιόν οπότε τώρα εργαζόμαστε σε θέματα βελτίωσης, ε, προσαρμογής ε, και έτσι είναι ρεαλιστικό και το χρονοδιάγραμμά μας το οποίο είναι το εξής τροπολογίες μέχρι τις 26 Μαρτίου 2 το μεσημέρι για να τις δημοσιεύσουμε πριν από το Πάσχα Εξέταση των τροπολογίων 23 Απριλίου και ψηφοφορία στις 16 Μαΐου. Οπότε, σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα, περνάμε στο επόμενο θέμα. Κοινή συζήτηση των τριών γνωμοδοτήσεων για την απαλλαγή. Η συγγήτρια είναι και η Swinburne. Ε, πρέπει να βιαστείτε λίγο γιατί η διερμηνία θα τελειώσει και μισή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να σας μιλήσω και για τη τρέση. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια. Και είχαμε την αρχική ανταλλαγή απόψεων και πρέπει να σας πω ότι αυτές οι τρεις απαλλαγές δεν θα πρέπει να μπουν στο ίδιο καλάθι με την αξιολόγηση του ΕΣΑ. Πάρα πολλέ από τις τροπολογίες είναι σε αυτό το πνεύμα. Λέμε τώρα για τρεις διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά υπάρχει ένα κοινό παρανομαστής στις τροπολογίες. Άρα, για να δούμε μερικά άλλα θέματα. Πολλέ αυτές τις τροπολογίες εξετάζουν το τι ρόλο έχουν πέσει αυτέ οι υπηρεσίε μετά την κρίση να υπάρχει σύγκληση εποπτείας, να υπάρχει και προστασία καταναλωτών. Σωστό, σωστό αυτό ήταν και για την ΕΣΑ. Ο Μπούσουλας και πρέπει να συνεχιστεί αυτό επίσης. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη προοικοδότηση για να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε να αποφασίσουμε επί τη βάση του ότι θα πρέπει εσωτερικά να καλυφθούν αυτά τα οποία ζητούν. Επίσης χρειάζεται ε, καλή οργάνωση και καλή δικαιολόγηση αύξηση σπόρων όπως είπε ο κύριος Γκίγκολτ και η κυρία Κάπελ στις ε, τροπολογίες. Και σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να ενημερωθούν αυτοί που αποφασίζουν για την πολιτική και έχουμε και τροπολογία Παπαδημούλη που λέει για τακτή αξιολόγηση. Επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και από την άλλη μεριά των εθνικών ομολόγων τους και σε διεθνές επίπεδο επίσης με ε, βιομηχανία. Επίσης ο κύριος Μαν είπε ότι θα πρέπει όλα αυτά να έχουν θεμέλιο την εμπιστοσύνη και ο κύριος Βέγκας το ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εξαρτησία των ε, φόρεων. Πολύ διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας. Κάποιες άλλες προτάσεις λένε θα πρέπει να, για τους καταγγέλους να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Μα ήδη έχουν λάβει τις πρωτοβουλίες αυτές ή υπηρεσίες πρόσφατα. Έχουμε και άλλες ε, επικοδομητικές προτάσεις. Μετάδοση στο ίντερνετ συναντήσεων, προσβασιμότητα στα έγγραφα, διαφάνεια για τα θεσμικά όργανα, αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλα αυτά αποτελούν προσθέμενη αξία στο κείμενο και για τις τρεις απαλλαγές. Λέμε ότι θα πρέπει να τηρούν την εντολή τους αυτές οι υπηρεσίες, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Να μην ε, επιχειρούνται αλλαγές πρώτου επίπεδου για διεύρυνση εντολής. Λάγκεν και Μαν, σωστές οι τροπολογίες για τη δική, σχέση με τη δική τους έκθεση για όποτε υπάρχει κάποια παρέκβαση από αυτές τις υπηρεσίες. Και πριν καλύψουμε τέτοιου είδους ισχυρισμούς στην απαλλαγή, ας το ψάξουν περισσότερο αυτό το θέμα των παρεκβάσεων. Μπάς και μπορούμε άλλη λύση. Και να ζητήσουμε από κάποια μονάδα πολιτικής να το δει το θέμα από πλευρά της Ευχαριστώ όλους τους σκιώδης ηγητές. Ευχαριστώ για τις προτάσεις τις συμβαστικές. Τις εγώ διανύμε. Ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Πιέζει ο χρόνος γιατί έχουμε ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και το λόγο στον κύριο Μαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΙ. Πολύ καλή δουλειά και πολλές καλές τροπολογίες. Χρειάζεται αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων της τραπεζικής αρχής για να δούμε και το κόστος του Brexit βεβαίως και της μετακόμισης. Είπε και η ότι πρέπει ο καθένας να μείνει στα πλαίσια της εντολής του, σωστό, καμία διεύρυνση και βεβαίως μεγάλη σημασία έχει και η αναλογικότητα και αυτό φαίνεται στη συμβαστική λύση που προτείνει ο ρόλος της CBA για την ενίσχυση των διεθνών εποπτικών δομών είναι πολύ σημαντική γραμμίζουμε ακριβώς την υποχρέωση ενημέρωσης της CBA και πρόσβασης ε, στα έγγραφα και συμφωνώ απολύτως. Για το θέμα ΕΙΟΠΑ και προστασίας των καταναλωτών ε, πάρα πολύ σημαντικό έχουμε βεβαίω και το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο πέρσι τον Δεκέμβριο εξέτασε την ΕΙΟΠΑ και είχε μια ξεκάθαρη θέση ναι όλα ήταν σωστά και νόμιμα ε, πρέπει να δούμε ακριβώς ε, και την κατανομή του προπολογισμού του 40% από τον κοινοτικό προπολογισμό 60% άμεσες εισφορές των κρατών μέλων πώς θα πρέπει να μειωθεί αυτό προσεχώς και βεβαίω έχουμε υποβάλει μια τροπολογία και ελπίζω να συμφωνήσεις υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα η ΑΙΟΠΑ να τηρήσει ε, κάποια βασικά πράγματα, εφαρμογή του πρωτογενούς δικαίου και τίποτα περισσότερο. Τρίτον, για την ΕΣΜΑ, σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κανένα πρόβλημα. Για τις άλλες αρμοδιότητες τώρα πρέπει να υπάρχει μια λογική αντιμετώπιση, να δημιουργηθούν κίνητρα για τους επενδυτές, ε, για την καταρξή της αγοράς οπωσδήποτε πρέπει η ΕΣΜΑ να το βλέπει και σίγουρα μια καλύτερη δικτύωση και βεβαίως να ενισχύσουμε την ένωση των κεφαλαίων Αυτά όμως σταδιακά και νομίζω ότι συμφωνώ. Έχουμε μια πολύ καλή κοινή θέση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπαγιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ναι, για τη δουλειά. Να θυμίσω την ε, σημασία για εμάς των, δύο αυτών, των τριών αυτών αρχών ώστε να έχουμε καλύτερο έλεγχο και διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γι' αυτό υποβάλλουμε μια σειρά από τροπολογίες που υπογράφουν την σημασία του, της αρμοδιότητας των τριών αυτών αρχών για μας είναι ουσιαστικότατο να έχουν τα απαραίτητα μέσα στη θέση τους όχι μόνο να έχουν την εντολή, να έχουν και τα μέσα για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους τα ανέφερε η συγγήτρια, η διαφάνεια, η προτεραιότητα στην προστασία των καταναλωτών, επ' αυτόν ε, συμφωνούμε και για τις τρεις αρχές είναι σημαντικό να έχουν μια ασφαλή δίωδο για τις καταγγελίες που θα μπορούσαν να υποβάλλονται από συγκεκριμένου ανθρώπους ε, για οποιαδήποτε παραβίαση, απάτη κτλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν ε, σταματήσουν οι διερμηνείς, κάτι μονανόημα νόημα να συνεχίσω αγγλικά πολλά από αυτά τα οποία θέλω να πω, τα έχουν πει οι συνάδελφοι. Ξετάζουμε λοιπόν αυτές τις εποπτικές αρχές ε, με την τρέχουσα μορφή τους. Ξέρουμε βεβαίως ότι αυτή ανακαθορίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ήδη υπόθηκε, σημασία έχει ακριβώς ε, να ενισχυθεί η συνοχή όπως είπε και η Σκοτ Κέιτο. Πρώτος στόχος, έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε και γι' αυτό ακριβώ πρότεινε η Κομισιόν κάποιες αλλαγές. Όσον αφορά το προϋπολογισμό και το ε, εσωτερικό τους κανονισμό, Νομίζω ότι ουσιαστικά έχουν εργαστεί πάρα πολύ καλά και οι μεταφορές είναι κάτω του επιτρεπόμενου ορίου. Τώρα, συμβάσεις ε, εκεί όπου κατά κανόνα υπάρχει ένα πρόβλημα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ε, εδώ πέρα στις συγκεκριμένες εποπτικές ε, αρχές ε, κανένα ζήτημα. Παρόλα αυτά η EBA σε κάποια stress test έβγαλε αποτελέσματα τα οποία αμέσως μετά αποδείχθηκαν λανθασμένα. Ενώ η ΕΙΟΠΑ στην εφαρμογή της οδηγίας για τη φεραγιότητα 2 οπωσδήποτε δεν πέτυχε την απαραίτητη σύγκληση. Οπότε νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν εδώ πέρα είναι δικαιολογημένη. Τώρα για την μετακόμιση στο Παρίσι μετά τον Brexit υπάρχει κόστος. Δεν ξέρουμε ακόμα σήμερα το ποιο θα είναι αυτό και ποιος θα το πληρώσει. Ελπίζουμε λοιπόν οι διαπραγματεύσεις του Μισελ Μπαναργιέ με τη Βρετανική κυβέρνηση να οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Συνολικά μπορώ να πω λοιπόν όσον αφορά τις διάφορες ε, τροπολογίες που σχολίασε η Κέιν Σουίνμπερν ε, είναι πάρα πολύ σωστές πηγαίνουν σωστή κατεύθυνση θεωρούμε ότι ε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και βεβαίως είμαστε και υπέρ της αρχής της αναλογικότητας δεν μπορεί για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια να δυσκολέψουμε την δουλειά των υπηρεσιών αυτών και να έχουμε περισσότερο διοικητικό βάρος. Ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Σουίμπορ για τη δουλειά που έχει κάνει και με τις τρεις γνωμοδοτήσεις. Από την πλευρά της ομάδας μας είναι γνωστό ότι έχουμε ενστάσεις για το συνολικό σχεδιασμό αυτού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ε, με βάση και αυτές τις ενστάσεις και σε ένα επικοδομητικό πνεύμα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την αποτελεσματική λογοδοσία και την εξασφάλιση μετρήσιμων αποτελεσμάτων από τη δουλειά αυτών των τριών θεσμών. Θεωρούμε σημαντικό ε, να υπάρχει μια τακτική και αναλυτική αξιολόγηση που θα βελτιώνει την κατανομή και την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Ε, όταν υπάρχουν πρόσθετα καθήκοντα και φόρτος εργασίας, αυτό να αντανακλάται με έναν αξιόπιστο τρόπο και στον προϋπολογισμό. Έτσι θα ενισχύσουμε και την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία αυτών των θεσμών. Θεωρώ επίσης απαραίτητο να συμμορφωθούμε αυτή η θεσμή με τα συμπεράσματα της ειδική έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επίσης είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνεργασία αυτών των τριών θεσμών και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, ε, νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας αναφορικά με τις συναντήσεις αυτών των θεσμών με ομάδες συμφερόντων και παράλληλα η ενίσχυση της προστασίας των καταγγελτών δημοσίου συμφέροντος. Ε, χαίρομαι γιατί η συγκήτρια έχει μια επικοδομητική στάση απέναντι σε κάποιες τροπολογίες που έχω καταθέσει και με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Thank you. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και δίνω λόγο στον κύριο Γκίκολτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Σουίντον για τα όσα έκανε για τις προσπάθειες συμβασμού... σε ένα κείμενο ήδη αξιόλογο. Κατά κάποιο τρόπο προτιμούμε το σχεδό κειμένο από το συμβαστικό κείμενο. Και υπάρχει και ένα θέμα το πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στην Επιτροπή μας. Εμείς φτιάξαμε τα έσας και προσδώσαμε εκεί μία εντολή η ισχυρότατη. Και εσείς κύριε Μάν το αποφασίσατε. Όπως και εγώ. Και όλοι, όλοι. Όλοι μας συμφωνήσαμε. Τώρα η ΕΣΑ ακριβώς προχωρούν πάνω σε αυτό το μονοπάτι αλλά κανένας δεν μπορούσε μέχρι τώρα να αποδείξει ότι υπήρχε κάποια παρέκβαση από την εντολή. Εμείς ε, είπαμε ότι εξασφαλίζουμε τώρα να είναι να υπάρχει λογοδοσία στο κοινοβούλιο. Ναι, όχι, δεν μου αρέσουν Δημήτρη και εμένα κάποιε πράξει των ΕΣΑ. Αλλά δεν έχω λόγου να πω ότι δεν ήρθαν εδώ, δεν του καλέσαμε, δεν απαντήσει κάποιε ερωτήσει. Μα αυτό έχει γίνει πολλέ φορέ και με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο. Αυτοί πάντοτε ανταποκρίνονται. Έρχονται μάλιστα και σε συναντήσει ε, σκιωδών εισηγητών και στέλνουν τους επικεφαλείς. Άρα επομένως ε, ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή τον έχουν ευξημένη υποχρέωση λογοδοσίας. Επίσης διέπονται από διαφάνεια όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε μήνα μας ενημερώνουν. Έχουμε συναντήσει συντονισμού για αυτά τα technical standards. Οπότε δυστυχώς τώρα έχουμε φτάσει σε κάποιες ε, συμβαστικές προτάσεις. Εκεί υπάρχει διατύπωση με κάποιους ισχυρισμούς ότι έχουν παραβεί την εντόλή τους. Ο ισχυρισμοί ότι θέλαμε να μας αναφέρουν σε τακτά διαστήματα όπως ε, στο συμβασμό ε. Μα το κάνουν αυτό, ήδη το κάνουν. Οπότε σας παρακαλώ μην ε, καλύψουμε τέτοιους χειρισμούς στην έκθεση. Για κλείστε, κλείστε, θα φύγουν οι διερμηνεί, λέει ο κ. Έτσι κι αλλιώ, έτσι κι αλλιώ, αγγλικά τα λέει, ο κύριο Γκίγκουλ. Ναι, αλλά θα πρέπει να κάνουμε την συνεδρίαση με την λέει ο κύριο Γκουαλτιέρη. Καλά, καλά, κλείνω. Οπότε σα παρακαλώ, όλα όσα έχουν σχέση με αυτού του ισχυρισμού να ψηφιστούν χωριστά. Εμεί θα καταψηφίσουμε του ισχυρισμού. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο, γιατί ζητήσατε από το Policy Department να τσεκάρει αυτού του ισχυρισμού. Άρα, όλα αυτά να στο policy department. Και εμείς, εμείς έναν προς έναν ισχυρισμό θα τον ε, γκρεμίσουμε ότι όλα αυτά έχουν έρισμα στον κανονισμό που διέπει τα ΕΣΑ. Τόμας, στείλε μου ό,τι έχεις για τέτοια παράβαση εντολής. Στείλ μου και εγώ θα σου βρω στον κανονισμό που δικαιολογείται. Ε, δεν θα πρέπει το κοινοβούλιο να είναι